Okay, people can start taking their seats now, colleagues. Παρακαλώ, καθίστε σιγά σιγά για να ξεκινήσουμε. Ο συνήθως με μικρή καθυστέρηση. Αλλά αν καθίσετε αμέσως θα την περιορίσουμε την καθυστέρηση. Είναι έκτακτη η συνεδρίαση αυτή, δεν είχε προγραμματιστεί από την αρχή του έτους, αλλά πολύ σημαντική παρόλα αυτά, γιατί προβλέπει διαρθρωμένο διάλογο με δύο επιτρόπους. Καταρχήν να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη με τρία σημεία, ή μάλλον τέσσερα. Το πρώτο είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Συμφωνείτε με την έγκριση του σχέδιου ημερήσιας διάταξης. Λαμπρά Σημείο 2. Ανακοινώσεις. Δεν υπάρχουν. Να σας υπενθυμίσω και την έκτακτη συνεδρία σήμερα στο στο Στρασβούργο στις 15 Μαΐου το απόγευμα. Ελπίζοντας ότι θα συνεχιστεί η πρόοδος ε, για τη συνένεση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Θα σας ενημερώσουμε εν καιρό. Ε, για να γράψετε στην ατζέντα σα την έκτακτη συνεδρίαση τη 15 η Μαου στο Στρασβούργο. Και περνάμε στο σημείο 3, διαρθρωμένο διάλογο επί του, σχεδίου εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο πρώτο διάλογο είναι με τον Επίτροπο Νέβεν Μίμιτσα, πολύ οικείο πρόσωπο φίλος της Επιτροπής μας. Και μετά την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Μίμητσα θα έχουμε το δεύτερο διαδρομένο διάλογο με τον Επίτροπο Στυλιανίδη. Ο διαδρομένος διάλογος είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είναι η ευκαιρία μας να επηρεάσουμε το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επόμενα χρόνια. Να ε, κοινοποιήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ε, προτεραιότητές μας και τις προσδοκίες μας από την τελευταία διετία αυτής της ε, κοινοβουλευτικής μας θητείας. Μερικοί όπως και εγώ φαντάζομαι δεν θα είμαστε στο νέο κοινοβούλιο και μετά τον Brexit. Άλλοι θα παραμείνουν. Οπότε είναι καλή ευκαιρία σήμερα να προωθήσουμε τις προτεραιότητές μας μέχρι το τέλος της ε, κοινοβουλευτικής μας θητείας και να προωθήσουμε και για το μέλλον την εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Ευχαριστώ θερμά τον Επίτροπο Μίμητσα που θα μας παρουσιάσει τις σκέψεις του, τις προβλέψεις του. Είναι πολύ σημαντική στιγμή για την αναπτυξιακή πολιτική με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τη Σύνοδο Κορυφής του Παρισιού. Έχουμε την αναδιάβαση αναθεώρηση για τα εξωτερικά μέσα χρηματοδότησης. Ξεκινήσαμε τριμερείς διαλόγους ε, για το FST. Ε, είναι καιρή αλλαγών και θα μας πείτε και τις δικές σας απόψεις για το τι προβλέπετε για την περαιτέρω πρόοδο και ευχαριστούμε που ήρθατε και το Γενικό Διευθυντή σας επίσης. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Είναι πάντα χαρά μου να έρχομαι για τον τρίτο διαρθρωμένο διάλογο φέτος για το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ξεκινήσω με λίγα λόγια για το συνολικό πλαίσιο πολιτικής που προτείνουμε και εκπονούμε από κοινού με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να καταλήξουμε στην Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη. Και μάλιστα τη στιγμή που η αξία της πολυμέρειας και της αλληλεγγύης αμφισβητούνται δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερη απόκριση και αντίδραση από, μια από ένα φιλόδοξο συλλογικό όραμα για την αναπτυξιακή πολιτική για να διατρανώσουμε και να επιβεβαιώσουμε τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα αυτά. Και η δική σας ε, συνεισφορά ήταν ζωτική σημασία για τη διαμόρφωση αυτού του νέου οράματος. Θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω όλους σας ε, και την Πρόεδρο, τους ε, συνεισηγητές Βέντα και Μόισε, καθώς και τους κοιόδης για την αφοσίωσή τους και την ε, επικοδομητική στράτευσή τους σε αυτή τη διαδικασία. Ε, Γενικώ, χάρη στην ε, ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταλήξαμε σε ένα κείμενο που ανταποκρίνεται στο υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών που είχαμε θέσει. Και μάλιστα δώσαμε ακόμη μεγαλύτερη έφαση στο γεγονός ότι η εξάλληψη της φτώχειας εξακολουθεί να παραμένει ύψητη προτεραιότητα και πρωταρχικό στόχος της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Επίσης, επισημάναμε τη σημασία που έχει η αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και η συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη. Ε, ενισχύσαμε και τη διατύπωση για την κοινωνία των πολιτών, ε, τα συστήματα υγείας, ε, ασφάλεια των τροφίμων, φορολογία και καλύτερα, θα σταθμίσαμε καλύτερα το, την ορολογία που χρησιμοποιούμε για τη μετανάστευση. Και στα πλαίσια του θεσμικού διαλόγου εξετάσαμε πολύ ε, σημαντικά απαιτητικά θέματα, όπω είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα καταπιστευματικά ταμεία, την ασφάλεια, την γεωργία και τη συστηματική παρακολούθηση των δεσμεύσεών μα για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Και από αυτή την άποψη, η νέα συνένεση θα πρέπει να βρει, να βρει τη σωστή ισορροπία ε, μεταξύ των απόψεων όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Πάντω, ε, ευελπιστώ ότι με αυτό το στόχο κατά νου θα βρούμε από κοινού κάποιους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε κάποια εκρεμή σημεία τις επόμενες μέρες και έχουμε πλησιάσει στην συμφωνία για το τελικό κείμενο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πόσο σημαντικό επίτευγμα θα είναι αυτή η συνένεση. Το να επιτρέψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σημαντικό παγκόσμιο φορέα να παρουσιάσει μια συνολική και περιεκτική προσέγγιση για την ανάπτυξη για να ανταποκριθεί στο πρόγραμμά της για το 2030 και μάλιστα με συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών. Ταυτόχρονα χαιρετίζω την θετική συνεισφορά σας ε, και μέσω του εισηγητού Μόιζε στη συζήτηση για τις μελλοντικέ μας σχέσεις με τις χώρες Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού και οι προτάσει μα ευθυγραμμίζονται πολύ με το δικό σα ψήφισμα και αποτελούν καλή βάση για την περαιτέρω συζήτηση. Βέβαια, βρισκόμαστε σε πρόωρα ακόμη στάδιο των συζητήσεων με τα κράτη-μέλη και υπάρχουν ακόμη κάποιες διαφορές απόψεων. Αλλά πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συνεννόηση προκειμένου να προτείνουμε κάποιες συστάσεις και για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και μάλιστα μέχρι το φθινόπωρο. Ταυτόχρονα Έχουμε επαφές με τις χώρες της Αφρικής, Καραβικής και Ειρηνικού και τις περιφερειακές οργανώσεις. Στόχος μου είναι να, συνεχίσουμε, να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μαζί τους ε, του χρόνου το καλοκαίρι επί τη βάση μιας ε, σχετικά κοινή προσέγγιση και οράματος. Και μάλιστα ο Λουί Μισελ και ο Πασκάλ Λαμή, πρώην ε, επίτροποι, συμβάλλουν στην διαμόρφωση της προσέγγισής μας υψηλότατο ε, πολιτικό επίπεδο στις ε, ενδιαφερόμενες χώρες και περιοχές. Και προσβλέπω στη δέσμευση και των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων, ώστε να μεταφέρουν τη συζήτηση αυτή στις ε, πρωτεύουσε και στις περιφέρειες, ώστε να αναβαθμιστεί η πολιτική διάσταση της μελλοντική συμφωνίας. Από πλευράς χωρών και, θέλουμε μία ομάδα αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για να ε, καθοδηγήσει, κατευθύνει βασικά τη διαδικασία, προκειμένου να επιτύχουμε την πρόοδο αυτή και να συνεχίσουν φυσικά τη δέσμευσή του καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία. Όπω ξέρετε, το 2017 θα είναι εξαιρετικά σημαντική χρονιά για τι σχέσει μα με την Αφρική, με τι ε, συνόδου κορυφή G7 και G20 και την πέμπτη Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Αμπιτζάν που θα γίνει, Αφρικής που θα γίνει στην Αμπιτζάν τον Νοέμβριο. Και μάλιστα θα υιοθετήσουμε κοινή ανακοίνωση με βάση τη συζήτησή μα για την αναζωογόνηση τη εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική. Η ανακοίνωση θα προτείνει μία ισχυρότερη, βαθύτερη εταιρική σχέση προσανατολισμένη στις δράσει για μεγαλύτερη σταθερότητα και ευημερία των δύο υπήρων. Στόχο είναι η δημιουργία θέσεων απασχόληση, κυρίω για του νέου και τι γυναίκε, αυξάνοντα ταυτόχρονα και τι επενδύσει, δημιουργώντα δηλαδή τι πρόσφορε συνθήκε ε, για τους επιχειρηματίες, ε, για την καινοτομία, για την επιχειρηματικότητα, κυρίως για ε, τομείς με ε, ψηλό δυναμικό δημιουργία θέσεων Απασχόληση, εξασφαλίζοντα οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Άλλο άξονα εργασιών είναι περισσότερο ανθεκτικέ κοινωνίε και κράτη, κάτι που προποθέτει ανανεωμένη δέσμευση των Αφρικανικών χωρών υπέρ τη ασφάλεια και τη ειρήνη. Ε, με δημοκρατικέ κυβερνήσει που θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλύτερη διαχείριση τη κινητικότητα και της μετανάστευση. Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική έχουν πολλά να κερδίσουν από ενισχυμένους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς, αλλά θα έχουν πολλά και να χάσουν αν αποτύχουμε στην ανάληψη αυτών των δράσεων. Γι' αυτό και περιμένω με αδημονία τις δικές σας προτάσεις για το πώς θα εξασφαλίσουμε μια αίσια διεκπαιρέωση της Συνόδου και γενικώ ε, καλύτερες σχέσεις με την Αφρική ένα συγκεκριμένο επίτευγμα που περιμένουμε από τη Σύνοδο Κορυφή ε, και αφορά τι ευρύτερε μα φιλοδοξίε είναι το νέο εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο. Πρόθεσή μα, ιδιαίτερα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη σχετική εγγύηση, είναι να ξεπεράσουμε τα υπάρχοντα μέσα και τις υπάρχουσες επενδυτικές δυνατότητες. Θέλουμε να στηρίξουμε ε, καινοτόμα μοντέλα χρηματοδότησης μέσω κάποιων χρηματοδοτικών ε, θεσμών και να ενθαρρύνουμε μεγαλύτερη ανάμειξη του ιδιωτικού κλάδου σε πιο ρηψοκίνδυνες επενδύσεις και κυρίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες και έφραυστες χώρες. Ε, και εκεί θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο όπως κοινωνικές και οικονομικές υποδομές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγαλύτερε μεγαλύτερες και ευκαιρίες για τις γυναίκες και τους νέους. Πρέπει να στηρίξουμε τις επενδύσεις, γιατί από μόνες αγορές δεν θα τα καταφέρουν να το κάνουν. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε την προσθετικότητα, που είναι κέρια έννοια για μας, που σημαίνει να επενδύουμε σε προγράμματα που θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο, σε περιοχές που χρήζουν ανάπτυξης, και για επενδύσεις που δεν θα υλοποιούνται χωρίς τη δική μας υποστήριξη. Δεν πρόκειται για ένα νέο μέσο ή εργαλείο, αλλά πρόθεση ενός μελλοντικού μοντέλου για βιώσιμη ανάπτυξη που θα ευθυγραμμίζεται με τις ε, διεθνείς μας ε, δεσμεύσεις και θα είναι εξίσου φιλόδοξο. Συνεχίζονται οι τριμερείς διάλογοι γιατί τον κανονισμό σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης που θα ευοδοθούν ε, προκειμένου να, να εγκριθεί ο κανονισμός πριν τις θερινές διακοπές. Και εδώ προσβλέπω στη συνεχή σα υποστήριξη ότι το επενδυτικό σχέδιο να γίνει λειτουργικό μέχρι το φθινόπωρο. Πέραν των επενδύσεων, η ισότητα των φύλων εξακολουθεί να αποτελεί ύψη προτεραιότητα των ε, ε, στόχων μας. Και επίσης ε, θα είναι γενικό στρατηγικό πλαίσιο για να χειραφετήσουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον πλανήτη. Και μάλιστα πρόκειται να δημοσιεύσουμε την πρώτη ετήσια μας έκθεση για την εφαρμογή του σχεδίου δράση για την ισότητα των φύλων και περιμένουμε θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την νοοτροπία ε, επιτόπου και μάλιστα εκατοντάδες οργανώσεις έχουν υποβάλει εκθέσεις και πάνω από 40 αντιπροσωπείες έχουν προετοιμάσει νέα ανάλυση για την ισότητα των φύλων προκειμένου να τη συμπεριλάβουν στον προγραμματισμό τους. Η ικανότητα του προσωπικού και η ε, πολιτική, ο πολιτικός ηγετικός ρόλος έχει βελτιωθεί ενισχύοντας τις ικανότητες ειδικευμένου και μη προσωπικού στα διάφορα γραφεία μας στο εξωτερικό. Επίσης, έχουμε φιλόδοξο στόχο να συμπεριλάβουμε δράσεις και να σε εκτιμήσουμε το φύλλο σε όλες τις νέες μας πρωτοβουλίες μέχρι το 2020. Περίπου 58% το, των πρωτοβουλειών μας πάνω των 9 δισεκατομμυρίων για το 2016 κατά σε μεγάλο βαθμό συνέβαλαν στην ισότητα των φύλων σε σχέση με το 43% που ήταν το ποσοστό για το 2015. Πέραν τη αύξηση τη χρηματοδότηση μέσω της, ε, του εξορθολογισμού των δράσεων και τη ανεκτήμηση τη ισότητα των φύλων, θέλουμε ειδικά κονδύλια για την ισότητα των φύλων που θα πρέπει να αυξάνονται και να χρηματοδοτούν πιο στοχευμένε δράσει, κυρίω για να γεφυρωθούν τα μεγάλα χάσματα στι χώρε εταίρου και να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, που είναι μια μάστιγα μεγάλων διαστάσεων που δεν γνωρίζει σύνορα, γενιές, κοινότητες ή κοινωνικές σφαίρες. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες για όλα τα κορίτσια και τις γυναίκες προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην παιδεία, την υγεία και τον οικογενειακό προγραμματισμό ε, τους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς πόρους και μια ηχηρή φωνή στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Χωρίς κάτι τέτοιο, η μάχη μας για την αηφόρο ανάπτυξη δεν θα στεφθεί με επιτυχία. Γι' αυτό καλώ όλους τους εταίρους μας να συνεργαστούν μαζί μα για την υλοποίηση αυτού του ζωτικού στόχου. Ένα άλλο τομέα με υψηλό δυναμικό ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων αναπασχόληση και που συμβάλλει στην εξάλληψη τη φτώχεια είναι ο ενεργειακό τομέα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τι χώρε εταίρου να αποδεσμεύσουν το τεράστιο φιλοπεριβαλλοντικό του δυναμικό, ε, δίνοντα πρόσβαση σε βιώσιμη και σε προσιτές ενέργεια προκειμένου να μειώσουμε το περιβαλλοντικό τίμημα του πλανήτη μας και των ε, επερχόμενων γενναιών. Και μέχρι το 2020 θέλουμε να δώσουμε πρόσβαση σε 40 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους ε, από τα 30 εκατομμύρια στην Αφρική και 15 εκατομμύρια ε, τόνους ισοδυνάμου διοξιδίου του άνθρακα και 11, τόνους, εκατομμύρια τόνους ισοδύναμα στην Αφρική και επίσης 5 γιγαβάτα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αφρική και 6,5 ε, στην ε, Ευρώπη. Και μάλιστα έχουμε δρομολογήσει 19 προγράμματα με γενικότερη επενδυτική δυνατότητα 4,8 δισεκατομμύρια για την ε, πρωτοβουλία ανανεώσιμη ενέργεια στην Αφρική. Κάτι που θα προσθέσει 1,8 γιγαβάτ ανανεώσιμη ενέργεια, που είναι περίπου 20% του συνολικού στόχου για την Αφρική. Προκειμένου να επιτύχουμε θα πρέπει να εμπλέξουμε όλους τους εταίρους μας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και αλλού, ακόμη και τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, άλλους χρηματοδοτικούς φορείς αλλά και την κοινωνία των πολιτών. Και γι' αυτό πρόσφατα συναντήθηκα με τον Επίτροπο Κανιέτε και με εκπροσώπους επιχειρήσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να συζητήσουμε επενδύσεις για την Αφρική και μάλιστα στις μέρες ανάπτυξης του Ιουνίου θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις προκειμένου να εμπλέξουμε τις χώρες εταίρους, χρηματοδοτικούς φορείς, ε, τον ιδιωτικό κλάδο και την κοινωνία των πολιτών. Έχουμε αναγνωρίσει ακόμη και στο πρόγραμμα για το 2030 και στις προτάσεις για τη νέα συνένεση ότι δεν θα έχουμε πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια και ειρήνη. Και στο πλαίσιο αυτό η πρόταση για την τροποποίηση του μέσου που συμβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη θα βοηθήσει ουσιαστικά τις χώρες εταίρους αλλά και τις περιφερειακές οργανώσεις να ε, αποτρέπουν όλο και περισσότερο και να διαχειρίζονται από μόνοι τους τις κρίσεις με κατάρτιση, συμβουλές και εξοπλισμό ε, σε εκτακτές συνθήκες. Και μάλιστα αυτό το μέσο μπορεί ήδη ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά δεν εμπίπτει στα κριτήρια αναπτυξιακής βοήθειας του ΩΣΑ. Και το το δραστηριοτήτων του 2015 ενέπιπτα στις δραστηριότητες αυτής της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας, την DAC. Βέβαια, οι νέες προτάσεις δεν θα αλλάξουν ε, ιδιαίτερα την, ε, την, ε, τις τάσεις αυτές, γιατί είναι μικρό το ποσό σχετικά, μόνο 100 εκατομμύρια που προσθέτονται στα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπει αυτό το εργαλείο που είναι 0,7 του ΑΕ. Επίσης δεν θα, δεν θα χρηματοδοτήσουμε αμυντικές δαπάνες ή αγορά πυρομαχικών και όπλων που συμβάλλουν μόνο στην μάχημη ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί η αγορα πυρομαχικων και οπλων που συμβαλλουν μονο στην μαχη ικανοτητα των στρατιωτικών φορέων γίνεται μόνο υπό, έκτακτε, υπό έκτακτους όρους όταν δεν υπάρχει δεν υπάρχουν πραγματικοί κρατικοί θεσμοί και με μόνο στόχο να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου. Και η δημιουργία δυνατοτήτων για την, αύξηση και την, για την ανάπτυξη και την ειρήνη θα πρέπει να συνάδει με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας. Όπως βλέπετε λοιπόν έχουμε ήδη προγραμματίσει το έργο μας για φέτος και του χρόνου. Και αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να προσδιορίσουμε και τις μελλοντικέ μας ε, πολιτικές και μέσα. Δεδομένων των προκλήσεων είναι σημαντικότερο από ποτέ η πολιτική μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη να προωθήσει ε, ένα πιο δίκαιο ε, και βιώσιμο κόσμο για όλους. Και θέλω να υπολογίζω στη δική σας εμπειρογνωμοσύνη και συνδρομή για την υλοποίηση των στόχων και περιμένω τις ερωτήσεις αλλά και τις προτάσεις για τα θέματα αυτά και σήμερα και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε. Πολλά πράγματα εξελίσσονται σε αυτή τη φάση. Βλέπουμε και στους τριμερούς διαλόγους, τριμερείς διαλόγους που είχαμε μαζί σας ότι οι εξελίξεις έχουν επιταχυνθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε μία ώρα το πολύ για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Μπόγκταν πρώτα και μετά η Ανελής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Θα ευχαριστήσω τον Επίτροπο Μίμητσα για την παρουσίασή του. Ελπίζω να κλείσουν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συνένεση για την ανάπτυξη. Η επιθυμία μας είναι να συνυπογραφεί την ε, ημερομηνία την εορταστική εν του Ευρωπαϊκού έτους για την ε, ανάπτυξη. Τώρα, το θέμα του συνδέσμου ανάμεσα στα θέματα ασφαλείας ε, και τη μετανάστευση και μετά από αυτά που συμβαίνουν και στην Τουρκία είναι σημαντικό για τη δική μου πολιτική ομάδα, αλλά νομίζω και για τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Το θέμα της κρίσης των προσφύγων θα παραμείνει στην επικαιρότητα για τα επόμενα χρόνια, από ό,τι φαίνεται. Σε ποιο βαθμό, λοιπόν, θα υπάρξει πραγματική εφαρμογή των προβλέψεων για την δημιουργία του καταπιστεύματος για την Αφρική τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να αντιμεταπιστούν οι βαθύτατες ε, αιτίες της ε, μετανάστευσης. Είναι ένα από τα θέματα αυτά λοιπόν. Το επόμενο θέμα, όπως είπατε ήδη, αναφέρομαι στην έκθεση Νόιζα για τις σχέσεις μετά την Κοτονού και μετά το 2020 μετά και έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις για τις νέες μορφές συνεργασίας. Εμείς είμαστε σαν ομάδα υπέρ μιας δεσπιστικής ε, πολιτικής συνεργασίας και ενός πολιτικού διαλόγου, αλλά και διαλόγου σε θέματα εμπορίου. Βλέπετε να γίνονται νέες εξελίξεις, να υπάρχουν νέες εξελίξεις όπως η περιφερικοποίηση, σαν παράδειγμα. αυτά. Ελπίζω να μπορέσουμε να συναντηθούμε κατά τη διάρκεια των ημερι... της ημερίδας για την ανάπτυξη. Άλλης, ευχαριστώ για τη συζήτηση που κάνουμε. Νομίζω ότι η καιροί είναι ιδιαίτερα ζωηροί και τίθεται το θέμα της έμφυλης προβληματικής και σε ποιο βαθμό όπως έχετε πει εσείς είναι κάτι το οποίο θα ληφθεί υπόψη. Εδώ θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Αναφερθήκατε και στα SDG. Υπάρχουν πέραν των SDG ε, και άλλα θέματα. Έχουμε μια έλλειψη, ενημέρωση στον τομέα των στόχων. Νομίζω ότι ακόμα και κάποιες πολιτικές ομάδες δεν είναι απόλυτα βέβαιες για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που κάπως διευκρινίσατε τα πράγματα. Αναφερθήκατε και για τα «και». Είχαμε εντατικέ συζητήσεις σε πολλά θέματα για την Κένια, την Μάλτα και εδώ έρχεται το θέμα των Panama Papers. Ήδη έχω αποστείλει μία επιστολή στην ομάδα των χωρών ΑΚΕ. Διαρωτώ με λοιπόν, υπάρχει ελπίδα να μετά από μια ενδιαφέρουσα ακρόαση που διοργανώσαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσουμε να συνδέσουμε το θέμα της ε, φοροδιαφυγής των Panama Papers με, την, ε, με τις πιστώσεις που δίδονται στη ΣΑΚΕ. Τώρα για την υποστήριξη συγκεκριμένων περιφερειών ε, και χωρών, στήριξη της Παλαιστίνης, στήριξη της UNCTAD είναι απαραίτητο και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επισκεφτούμε επιτέλους τη Γάζα. Σαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μας το επιτρέπουν. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στη λωρίδα της Γάζα, οπότε θα πρέπει να μπορέσουμε επιτέλους να πάμε. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την διάσκεψη την οποία διοργανώσαμε για την αλυσίδα προμηθειών στον τομέα των ενδυμάτων. Υπήρξαν άνω των 100 ΜΚΟ, το Κοινοβούλιο, εκπρόσωποι από την Ινδία, από το Μπαγκλαντές και νομίζω ότι εμείς σαν Κοινοβούλιο βλέπουμε ότι είναι θετικό το ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τη δέουσα επιμέλεια της, του ΟΣΑ θα ληφθούν υπόψη στον τομέα της ένδυσης από εδώ και πέρα. Γι' αυτό θα θέλαμε λοιπόν αν είναι δυνατόν να υπάρξει μια δεσμευτική λήψη υπόψη της δέουσας επιμέλειας. Και έτσι να μπορέσουμε να πάρουμε τις πρωτοβουλίες που αναφέραμε στην συνάντηση που είχαμε. Πολλές είναι οι χώρες που ενδιαφέρονται για το θέμα και θα θέλαμε να το υπογραμμίσουμε. Υπάρχει επίσης και το θέμα της, του μέσου για την ειρήνη και την ασφάλεια. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα το πρωί να δούμε πώς οι Γερμανοί το αντιμετωπίζουν. 200 ε, εκατομμύρια δίδουν, είναι ένα μικρό κομμάτι, αλλά η Γερμανία ε, πέρυσι διέθεσε 100 εκατομμύρια, φέτος 130 εκατομμύρια έχουν μια ξεχωριστή γραμμή στον προπολογισμό στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Δεν είναι θέμα να ληφθεί υπόψη το αν είναι συμβατό με τον ΤΑΚ ή όχι. Πάντως, εξ ονόματος πολλών μελών της ομάδας των σοσιαλιστών και των υπολείπων φίλων της Επιτροπής, να βγάλουμε τα DJI από το μέσο αλλά να λάβουμε υπόψη μας μια μακροπρόθεσμη λύση ε, για το επόμενο δημοσιονομικό, γιατί το θέμα της συμβατότητας με τα ΝΤΑΚ είναι καθοριστικό για μας. Νομίζω ότι το γερμανικό παράδειγμα θα πρέπει να ακολουθηθεί με ότι αυτό συνεπάγεται και νομίζω ότι ο πίνακας ο γερμανικός είναι πάρα πολύ κατα... κατατοπιστικός. Οι ΜΚΟ το ζητούν αυτό, οι εκκλησίες το ζητούν αυτό, το Γερμανικό Υπουργείο για την Ανάπτυξη το επιζητά αυτό. Δεν θέλουν να δούνε τμήματα του προϋπολογισμού ECI σε αυτό το κομμάτι. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία ήθελα να σας θέσω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σήμερα εδώ. Για τους φιλελεύθερους ο κύριος Βάρινεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Άνελιτς ε, ανέφερε όλα τα ζητήματα που είχα και εγώ στο μυαλό μου. Εδώ, στην Επιτροπή μας, ετοιμάζουμε μια γνωμοδότηση σχετικά με αυτό το μηχανισμό που συνεισφέρει, συμβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη και έχουμε πολλές ανησυχίες αναφορικά με τις επιπτώσεις αυτού του μηχανισμού στην ε, αναπτυξιακή πολιτική. Είναι μικρό, όμως υπάρχει η πιθανότητα μεγάλης αύξησης στο μέλλον. Η πιο ριζοσπαστική βέβαια ιδέα μόλις παρουσιάστηκε από τον Άνε Λίτς. Βασικά εγώ ως εισηγητής ήμουν έτοιμος να αποδεχθώ την πρόταση της Επιτροπής, τη δομή. Όμως πρέπει να έχουμε κάποιες ε, εγγύησει για τις ε, αναπτυξιακές πτυχές του χρηματοδοτικού μηχανισμού. Η πρόταση της Επιτροπής είναι πολύ περιορισμένη ε, όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής της, για ποιους σκοπούς είναι η χρηματοδότηση, πώς θα χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως. Εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή ΑΦΕΤ, έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης που θα αλλάξει την πρόταση της Επιτροπής ε, με έναν ριζοσπαστικό τρόπο. Η πιο ε, αλλαγή θα είναι στην ουσία η αλλαγή της δομής ε, στο άρθρο 3, όπου η Επιτροπή επι... προτείνει το ε, Α και β να είναι μια αρθριστική οντότητα, έτσι ώστε όλοι οι όροι στο α και β να πληρούνται. Στην ΑΦΕΤ ε, προτείνουν αντί για το end να βάλουμε or, αντί για το και να βάλουμε ή διαζευκτικό, ώστε ο μηχανισμός να χρησιμοποιείται μόνο όταν ε, οι όροι του τμήματος Β, της παραγράφου Β πληρούνται. Αυτές λοιπόν είναι οι προτάσεις της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Τώρα το Συμβούλιο έχει και αυτό καταθέσει τη θέση του. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν αν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο για τη θέση του Συμβουλίου. Δεύτερον, ελπίζω όταν γίνει η τριμερής διάλογος η Κομισιόν να, βασισ... να παραμεινθεί της βασικής ε, προληπτικής γραμμής που ακολουθεί. Γιατί το έγγραφο δεν είναι και πολύ κακό από τη δική μας άποψη τουλάχιστον. Συμφωνώ λοιπόν με αυτά που είπε ο Άνελίτς σχετικά με το χρηματοδοτικό μηχανισμό. Ευχαριστώ Μαρία Χόιμπουργκ. Ευχαριστώ Λίντα, ε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Ε, ήθελα να πω άλλο ένα ε, πράγμα για τις υπερεθνικές επιχειρήσεις, την απορρόφηση των κραδασμών, για την ε, ε, ανθρώπινα δικαιώματα και την παραβίασή τους. Υπάρχει μία μελέτη, αυτή εδώ που βλέπετε, σχετικά με τα όσα έγιναν στο επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έγινε πέρυσι. Έχει να κάνει με το land grabbing, τα ανθρώπινα δικαιώματα την αρπαγή γης γενικά ε, σε περιοχές που είχαν συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε συγκεκριμένα λοιπόν να δείτε τι συνέβη και σύμφωνα με τη μελέτη υπάρχουν πράγματα που δεν έχουμε δει. Τώρα για τη συνένεση ε, στη φάση των διαπραγματεύσεων που βρισκόμαστε έχουμε δει λίγο πολύ τι συμβαίνει. Ε, ε, στη Γερμανία λέμε ότι δεν μπορείς ε, να μιλάς για κάτι που δεν έχει ακόμα παρουσιαστεί μπροστά σου, δεν μπορείς να μιλάς για αυγά που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα, όπως λέει το ρητό μας. Ε, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τώρα που έχουμε αυτό το κείμενο για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνένεση από αυτού. Να μιλήσω όμως και άλλη μια φορά ξεκάθαρα και να πω ότι στη συζήτηση το Φεβρουάριο στο Στρασβούργο μιλήσαμε και αποφασίσαμε να έχουμε ε, μία συνένεση για την ανάπτυξη και όχι για την ασφάλεια και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Το τελευταίο θέμα είναι ένα θέμα κλειδί που δημιουργεί δυσκολίες ε, στην διαπραγμάτευση γιατί υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Εσωτερικά πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Και άλλο ένα θέμα στις ε, διαπραγματεύσεις είναι η εφαρμογή. Ε, πώς και πότε ε, και ποια μέτρα θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσους στόχους θα εφαρμόσει μέσα στα πλαίσια της συνένεσης. Σύμφωνα με τα όσα έχουμε τώρα, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα κάνουν αυτά που πρέπει σε 100, είναι 150 οι στόχοι και είναι πολύ σημαντικό η Κομισιόν να έχει ένα σχέδιο δράσης για όλα αυτά. Δεν πρέπει να αφαιθούμε χωρίς να έχουμε συγκεκριμένες δραστηριότητες για αυτές τις 150 προθέσεις μέσα σε ένα ρεαλιστικό χρονικό πλαίσιο πάντοτε. Περιμένω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έγινε και την τελευταία φορά στη συνένεση, γιατί, να υπάρχει ένα σχέδιο για την εφαρμογή, ένα staff planning document. Ε, έχουμε και για την ανθρωπιστική βοήθεια ένα τέτοιο έγγραφο εργασίας υπηρεσιακό, ε, έτσι ώστε να μπορούμε να εργαστούμε σωστά. Θα είναι καλό λοιπόν και για τη νέα συνένεση να έχουμε ένα αντίστοιχο έγγραφο για να μπορεί να εργαστεί το Κοινοβούλιο επί του τακτικού διαλόγου ε, βάσει αυτού του εγγράφου και να γίνουν και οι αντίστοιχες συνομιλίες βάσει αυτού. Τέλος, μια τελευταία ερώτηση. Ε, το περασμένο έτος, πέρυσι, είχαμε ως δράση για αυτό το έτος από την Επιτροπή ε, είχαμε ε, ζητήσει ε, ένα σχέδιο δράσης για την αρπαγή γης ε, στις χώρες εταίρους. Φαίνεται λοιπόν ότι παραμένει το πρόβλημα και πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα δράσουμε. Όταν κανείς εκδιώκεται από τη γη του, στην ουσία βρίσκεται σε φυγή, ακόμα και προς την Ευρώπη. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερα να δω ε, τι γίνεται με το σχέδιο δράσης κατά της αρπαγής ε, γης. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και άλλη μία ερώτηση για τον πρώτο γύρο, Γνάτσιο Κοράου. Και μετά θα κάνουμε ένα δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ, Λίντα. Καλησπέρα, Επίτροπε. Θα κάνω μία ερώτηση σχετικά με την εταιρική ευθύνη γιατί θεωρώ ότι πολλά από τα πράγματα από τους τομείς που αναφέρατε στην παρέμβασή σας σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο με, την, με τη δραστηριότητα των υπερεθνικών των πολυεθνικών θα λέγαμε επιχειρήσεων και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αποτελεσματική δράση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον τομέα της εταιρικής ευθύνης. Πρόσφατα στο Κοινοβούλιο αναγνωρίσαμε όλο ένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πολλές εκθέσεις σχετικά με την ε, εταιρική ευθύνη. Ξεκινώ, αλλά υπάρχει και ο τομέας της ένδυσης, πρώτες ύλες. Οι πολιτικές ομάδες ε, φαίνεται να συμμερίζονται το ίδιο όραμα προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για την Επιτροπή, γιατί ακόμα περιμένουμε μια απτή δράση από την πλευρά τους ως follow-up για τις ε, εκθέσεις που εμείς εγκρίναμε πέρυσι. Τον, στις 19 Ιουλίου του 2016 με μαυρία πλειοψηφία το Κοινοβούλιο ενέκρινε μία έκθεση πρωτοβουλίας, ήμουν εγώ ο εισηγητής, για την ευτερική ευθύνη και τις καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, ε, φαίνεται λοιπόν ότι αυτό η Κομισιόν δεν το έχει προχωρήσει. Δεύτερον, για τις ε, παγκόσμιες αλυσίδες αξίας είχαμε απόψεις ε, από όλες τις πολιτικές ομάδες που πηγαίναν προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό μας επέτρεψε να περιλάβουμε σχεδόν όλες τις τροπολογίες στις συμβαστικές τροπολογίες του πλαισίου για έναν συνεργατικό διάλογο είμαι σίγουρος ότι η γνωμοδότηση, η έκθεση που σχετίζεται με αυτή θα είναι ένας καλός τρόπος να θέσουμε έμφαση σε βασικές έννοιες και να έχουμε μετά απέτηση για αυτή εφαρμογή αυτού που απαιτήσαμε ε, τον Οκτώβρη. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα θετικό κλίμα από όλες τις πολιτικές ομάδες ε, που είναι σπάνια θα έλεγα, δυστυχώς πρέπει να κάνω ένα αρνητικό σχόλιο από τη μία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλο και περισσότερο εμπλέκεται σε αυτό το θέμα και γίνεται πιο ενεργό. Οι πολιτικές ομάδες συνεργάζονται περισσότερο, όμως η Κομισιόν συνεχίζει να αγνοεί τη φωνή μας και να αντιτίθεται στο όραμα του Κοινοβουλίου. Πάνω από μία φορές σε αυτό το κοινοβούλιο είδαμε την Digitrade στην ουσία να αντιτίθεται στις δεσμευτικές, σε δεσμευτικούς κανόνες για αυτό το θέμα. Και έκανα και μια συγκεκριμένη ερώτηση και η Κομισιόν έδωσε μια πολύ έτσι φευγαλέα απάντηση. Γι' αυτό το λόγο σήμερα στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα ε, ζητήματα ελπίζοντας σε μια συγκεκριμένη απάντηση. Ξέρει η Κομισιόν ότι εγκρίθηκε η έκθεση με μεγάλη πλειοψηφία για να μπορέσει να αναλάβει δράση. Τώρα, έχετε σκοπό να, πάρετε, να αναλάβετε συγκεκριμένη δράση. Ε, για τα VGs επίσης, ε, ποιες είναι οι οι δράσεις που θα έχετε στις συγκεκριμένες ε, γενικές διευθύνσεις. Αυτό είναι ο πρώτος γύρος. Ε, κύριε Επίτροπε, θα μπορούσατε να απαντήσετε 10 λεπτά σε αυτόν και μετά να πάμε στον επόμενο γύρο. Ε, και μετά έχουμε 5-6 συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο. Πολύ ενδιαφέρον για αυτά που έχετε να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά για τα σχόλια, τις απόψεις, τις ερωτήσεις σας για πολλά και σημαντικά θέματα του προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και τις κατευθυντήριες γραμμές της αναπτυξιακής μας πολιτικής για το μέλλον. Να ξεκινήσω με το σύνδεσμο μεταξύ μετανάστευσης, ασφάλειας και ανάπτυξης. Είναι διτώ αυτό το θέμα. Όντως, θα πρέπει να βελτιώσουμε και να εξυγχρονίσουμε τους ισχύοντες μηχανισμούς και τα μέσα που έχουμε, ώστε να ανταποκριθούμε ε, στο γενικό ζήτημα των δεσμών της ασφάλειας με την ανάπτυξη, όπως γίνονται δεκτεί αυτή η θεσμή στο παγκόσμιο πρόγραμμα για την ανάπτυξη. Γιατί υπάρχει συσχετισμός και δεσμός. Και αυτό το έχουμε αναγνωρίσει και δεχτεί και στις δικές μας ε, συγκεκριμένες δράσεις. Γιατί η ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Και αν δείτε ε, στο θεματολόγιο της Νέας Υόρκης για το 2030, η στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη, διαπιστώνεται ότι η ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά εξετάζει πιο διασταλτικά τα μέσα και τους μηχανισμούς αναπτυξιακής βοήθειας. Θα πρέπει λοιπόν να εξυγχρονίσουμε τους μηχανισμούς που έχουμε και που συμβάλλουν στη σταθερότητα και στην ειρήνη, αλλά να κρατήσουμε ε, απαράβατη αυτή την κόκκινη γραμμή και δεν είναι να μην την υπερβούμε. Δηλαδή, η χρηματοδότηση από την ανάπτυξη ή από οποιαδήποτε άλλη δημοσιονομική γραμμή ε, να μην ε, αφιερώνονται σε χρηματοδότηση αμυντικών αναγκών ή στην αγορά όπλων και πυραμαχικών. Αυτή είναι η κοινή γραμμή που απορρέει και από τις συνθήκες σε καμία περίπτωση αναπτυξιακά κονδύλια να μην χρησιμοποιούνται για την κάλυψη στρατιωτικών ή αμυντικών αναγκών. Θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε, παραλαμβάνω, τα ισχύοντα μέσα, αλλά να κρατήσουμε υψηλό το επίπεδο των δεσμεύσεών μας και να αποφεύγουμε την κοινωτική χρηματοδότηση για στρατιωτικούς σκοπούς. Και στο μέλλον χρειαστούμε μια διαφορετική προσέγγιση σε, στις επιχειρήσεις που σήμερα χρηματοδοτούμε από τα αναπτυξιακά μας μέσα, όπως είναι η Άμισον. Θα μπορούσε να ενταχθεί στη μελλοντική μας ε, αμυντική πολιτική, στο μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκεί, στο επόμενο πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο θα συζητήσουμε, θα αναλύσουμε και θα συμφωνήσουμε για τη μακροπρόθεσμη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε, αυτές τις, σε αυτή τη συσχέτιση ασφάλειας και ανάπτυξης. αυτή τη, φορά, αυτή τη στιγμή έχουμε το μέσο για την ε, σταθερότητα και ειρήνη. Μέσω αυτού συμβάλλουμε στη σταθεροποίηση της εσωτερικής ασφάλειας σε χώρες εταίρους μας. Θα αναλύσουμε όλα, όλες τις περιπτώσεις και τα παραδείγματα που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε νέα ε, μέσα και μηχανισμούς, αλλά προς το παρόν θα ήθελα να επικεντρωθούμε στη συγκεκριμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. και αυτή, αυτή η πρόταση αποτελέσει τη βάση στην επόμενη νομοθετική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά το σύνδεσμο, το δεσμό μετανάστευσης και ανάπτυξης. Πολύ συχνά ακούμε τη, την άποψη ότι κάποια αναπτυξιακά κονδύλια θα αφιερωθούν για τη χρηματοδότηση στόχων που δεν είναι κατά παράδοση αναπτυξιακή αλλά θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της μετανάστευσης ή τη διαχείριση των συνόρων. Εγώ δεν θα έλεγα ότι η χρηματοδότηση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας ή των στόχων DAC που είναι συναφή με την ε, μετανάστευση δεν σημαίνει αυτόματη αφαίρεση κονδυλίων από τη χρηματοδότηση των γενικών αναπτυξιακών μας στόχων. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει φυσικά στενός δεσμός μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης, κάτι που έχει αναγνωριστεί και από το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και ελπίζω ότι θα αναγνωριστεί και στη νέα μας συνένεση για την ανάπτυξη. Αυτό άλλωστε αντικατοπτρίζεται και σε μια πλειάδα τομέων για πιθανή χρηματοδότηση αναπτυξιακή, η εξάλληψη της φτώχειας και η αντιμετώπιση των αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης ε, είναι, ε, είναι στόχοι που συμβαδίζουν, ε, για να μην πω ότι ταυτίζονται. Γιατί η εξάλληψη της φτώχειας είναι ο βασικός στόχος της αναπτυξιακής μας δράσης και η φτώχεια είναι μία από τις αιτίε της παράτυπης μετανάστευσης. Οπότε είναι σαφώς ελεύθερες αυτές οι δύο έννοιες μετανάστευση και ανάπτυξη. Επίσης, αυτά τα θέματα έχουν κάποια συνάφεια και με τις δράσεις μας για την πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροδιαφυ... φοροαποφυγής και φορολογικής απάτης ή τις προτάσεις για τη φορολογική βάση. Δεν θα ήθελα τώρα να προεξοφλήσω την έκβαση των συζητήσεων για τα έγγραφα του Παναμά. Δεν μπορώ να προβλέψω τις εξελίξεις εκεί. Χαίρομαι για τις πρωτοβουλίες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ειδική Επιτροπή και Επίσης, ε, περιμένουμε όλους τους φορείς που αναλύουν αυτό το θέμα να διεκπαιρεώσουν τις αναλύσεις τους. Πάντως, το έγγραφο του Παναμά, το σκάνδαλο αυτό ήταν ένα καλό παράδειγμα που μας δείχνει γιατί θα πρέπει να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή μας συνεργασία και στο τομέα της φορολογίας και να το κάνουμε και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στις χώρες εταίρους. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε και τους δικούς τους πόρους προς αυτή την κατεύθυνση. Γεγονό που συνάδει και με τις πρωτοβουλίες μας για την καλύτερη φοροείσπραξη και τις ε, καλύτερες δαπάνες. Πιο στοχευμένες δαπάνες, που είναι γενικότερο στόχος και της αναπτυξικής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά την ε, Παλαιστίνη, και την γενική μας ε, δέσμευση στην περιοχή. Η αναπτυξιακή βοήθεια και αναπτυξιακή συνεργασία στην Παλαιστίνη είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα κοινού προγραμματισμού και κοινών δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και των 21 κρατών μελών. Θα συνεχίσουμε να επηρεάζουμε θετικά την ανάπτυξη στην Παλαιστίνη, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά φαντάζομαι και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα συνεργαστούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συμβάλλει πλήρως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ενίσχυση και στη βελτίωση ε, της αναπτυξιακής μας συνεργασίας με την Παλαιστίνη. Συμπεριλαμβανομένης και της επίσκεψης αντιπροσωπείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λωρίδα της Γάζας. Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για την ένδυση, όντως ήταν πολύ καλή η συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα εκπονήσαμε και το έγγραφο εργασίας για την πρωτοβουλία αυτή για την ένδυση. Και θα πρέπει να ενισχύσουμε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας σε αυτό το σημαντικό τομέα βιομηχανικής δραστηριότητας. Η πρωτοβουλία για την ένδυση είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τις αλυσίδες αξίας και θα εξασφαλίσουμε το σεβασμό κάποιων προδιαγραφών ε, επισήμανσης, αλλά και το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διαδικασία παραγωγής ενδυμάτων. Επίσης, ε, θα θέλαμε στο έγγραφο εργασίας να προωθήσουμε αυτή την πρωτοβουλία και να μπορούμε εν καιρό να αξιολογήσουμε τον πραγματικό αντίκτυπο και την ε, αξία μιας τέτοιας προαιρετικής προσέγγισης γιατί δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα αυτή η πρωτοβουλία για την ένδυση. Και περιμένουμε τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να οδεύσουμε προς, μια πρόταση που θα είναι και νομικά δεσμευτική για τον τομέα της ένδυσης. Αλλά πρώτα θα πρέπει να εξερευνήσουμε πλήρως το δυναμικό της εθελοντικής προσέγγισης που έχουμε προτείνει στη δική μας πρωτοβουλία, στο έγγραφο εργασίας και μετά να δούμε αν θα οδεύσουμε και μια νομικά δεσμευτική πρόταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γενικότερο ζήτημα της εταιρικής ευθύνης, θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει επικοδομητικά στο έργο της Διακυβερνητικής Ομάδας των Ηνωμένων Εθνών που θα προτείνει ένα νομικά δεσμευτικό μέσο για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και χαίρομαι που στη σχετική ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών οι συζητήσεις καλύπτουν όλες τις ε, ε, επιχειρήσεις, όχι μόνο τις πολυεθνικές εταιρείες, αλλά όλες τις εταιρείες και χαιρόμαστε γιατί η συζήτηση είναι ανοιχτή και επικοδομητική. Και έχουν υποβληθεί πολλές ε, εύστοχες προτάσεις από τα μέλη της ομάδας. Βέβαια, το ζήτημα είναι περίπλοκο και μερικές φορές τεχνικό και άπτεται πολλών ε, θεμάτων. Γι' αυτό και περιμένουμε στα τέλη του έτους την επόμενη συνεδρίαση της διακυβερνητικής αυτής ομάδας εργασίας στο Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να συμβάλλουμε με τις δικές μας προτάσεις. Πάντως αυτό το θέμα ε, του συνδυασμού των επιχειρήσεων με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι προσφυλές. Ε, και αφορά όχι μόνο την εταιρική ευθύνη, αλλά και το θέμα της αρπαγής γεών. Πάντως θα συμβάλλουμε και εμείς ώστε να έρθει σε αίσιο πέρας η πρωτοβουλία, η σχετική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών. Also, some... Κάποια από τα θέματα τα οποία συνδέονται με την συνένεση. Η διαδικασία όπως έχω ήδη πει στην αρχική μου παρέμβαση η διαδικασία συμφωνίας για το κείμενο της συνένεσης έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά στο υιοθετήσουμε πρώτα και μετά ας προσπαθήσουμε να δούμε τον καλύτερο τρόπο για να εφαρμόσουμε την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ισχυρή ευθύνη εδώ. Πρέπει να κρατήσει το ρόλο τον οποίο έχει στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Και γι' αυτό η βασική προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει για να ασκηθεί η ευθύνη αυτή είναι ακριβώς εδώ αυτή η συνένεση. Η συνένεση αυτή, όπως είπα, είναι διαφορετική από ό,τι στο παρελθόν σε επίπεδο συνένεσης με την προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αλλαγή. Και οι μεμονωμένες χώρες και ε, οι εμπλεκόμενοι γενικότερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο, εκφράζουν τις προτεραιότητές τους, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν εξίσου υπόψη και από τα κράτη-μέλη και από το κομμάτι της ανάπτυξης που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι λοιπόν στην επόμενη φάση θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο πρόγραμμα δράσης ή έστω μια κοινή συμφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Επιτροπή για την εφαρμογή της συνένεσης για την ανάπτυξη. Νομίζω ότι έχω απαντήσει σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις. Καλώς περνάμε στον επόμενο γύρο. Μπορείτε να σκεφτείτε και να ελέγξετε. Πέντε ομιλητές τώρα, θα πρέπει τέσσερις και μισή να τελειώσουμε κύριε Επίτροπε. Θα έρθει ο επόμενος κύριος. Στυλιανίδης, ο κύριος Κόζα. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κυρία Κόζα, συγγνώμη. Να είμαι σύντομος. Έχω τρεις ερωτήσεις, εκ των οποίων οι δύο ήδη ε, αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους, άρα μου μένει η τρίτη ερώτηση. τα μέτρα εξέβρεσης θέσεων εργασίας, τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις γυναίκες και τα παιδιά αναφέρθηκαν. Αναφέρθηκε ότι δίνεται μεγάλη σημασία στην ισότητα των φύλων. Επίσης, στο κείμενο της Κομισιόν αναφέρονται αυτά τα ζητήματα και υπάρχει και μια έκθεση από το Κοινοβούλιο σχετικά. Εσείς πώς θέλετε να εφαρμόσετε όλα αυτά στην πράξη. Πρέπει να θυμάστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία ε, κυρώση, μία χάρτα των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, σχετικά με τα άτομα με αναπηρία. Πώς θα περάσει αυτό την εργασία μας εδώ και φυσικά την ισότητα των ε, γυναικών, των παιδιών και των ανθρώπων με αναπηρία. Όλα αυτά αναφέρονται. Ε, αυτό δεν το αναφέρω σε επίκριση. Απλώς ε, θα ήθελα μία υγιή πρόταση. για να μπορέσει να ληφθεί υπόψη και η πλευρά των ανθρώπων με αναπηρία. Αυτή είναι η συγκεκριμένη ερώτησή μου προς εσάς. Αν τελικά στην πράξη θα μπορέσουν αυτά ρεαλιστικά να εφαρμοστούν. Thank you. Um, Ευχαριστώ, Ερίκη Κεραίρο. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, δεν θα επαναλάβω λοιπόν θέματα τα οποία ήδη έχουν τεθεί να κάνω ορισμένα σχόλια και μια συγκεκριμένη ερώτηση όμως. Νομίζω ότι είναι σωστή ιδέα το να συνδέσουμε και τον Πασκαλαμή στο, στην επεξεργασία των θέσεων για την περίοδο μετά το Κοτονού. Η αναθεώρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και ταυτόχρονα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αξιολόγηση των επιπτώσεων στις δημοσιονομικές μας πολιτικές και κατά πόσον ε, επηρεάζονται όχι μόνο οι χώρες ΑΚΕ αλλά κυρίως οι χώρες ΑΚΕ βέβαια ε, στα πλαίσια του προγράμματος μετά το Κοτονού. Σχετικά με τη συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής να δούμε ε, πώς μπορούμε να διευρύνουμε λίγο το πρόγραμμα των επενδύσεων. Το πρόγραμμα αυτό ε, συγκεντρώνεται κυρίως σε κάποιες 7 ή 8 κατά προτεραιότητα χώρες, ενώ βασική μας ε, θα έλεγα προσδοκία, θα είναι φιλοδοξία, θα είναι να μπορέσουμε να επενδύσουμε σε πολύ περισσότερες χώρες. Λοιπόν, έχει, είναι καλή στιγμή για να θέσουμε το θέμα. Τρίτον, η τροποποίηση την οποία αναφέρατε για το μέσο ειρήνης και αλληλεγγύης. Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο χρονισμός τον οποίο προβλέπετε, γιατί στην Ολομέλεια των ΑΚΕ τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο προβλέπεται να εγκριθεί μια έκθεση πάνω στα θέματα της ασφάλειας και της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Εγώ είμαι από πλευράς των Ευρωπαίων ο εισηγητής θα πρέπει να προηγηθούν βέβαια συζητήσεις με την άλλη πλευρά, την Αφρικανική ή τις υπόλοιπες χώρες και η Τζουντίτ Αργεντίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία ερώτηση για τα ορυκτά από ζώνες συγκρούσεων. Πάει κάποιος καιρός που είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό Ήδη το είχαμε πρώτο συζητήσει το 2010 και ολοκληρώσαμε την ομοθετική διαδικασία πρόσφατα. Μαζί με την πρόταση την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δέουσα Επιμέλεια στον τομέα των ορεκτών αυτών, ήρθε και η υπόσχεση, θα έλεγα, για τα λεγόμενα συνοδευτικά μέτρα. Αυτό ήταν πάντα ένα τμήμα της αναπτυξιακής ευθύνης και όχι της εμπορικής ε, ε, ατζέντα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε η εφαρμογή σε μια χώρα όπως το Κονγκό να γίνεται με τον σωστό τρόπο. Ένα άλλο θέμα έχει σχέση με τις ερωτήσεις οι οποίες έχουν ήδη τεθεί για τον τομέα της φαντουργίας και της ένδυσης και τις δεσμευτικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Και εδώ χρησιμοποιούμε την ίδια μέθοδο η οποία χρησιμοποιήθηκε και για τα ορικτά από ζώνες συγκρούσεων. Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ για τον τομέα της ένδυσης θα πρέπει να εφαρμοστούν όπως γίνεται ήδη στην Ευρώπη σε θελοντική βάση. Δυστυχώς δεν γίνονται απόλυτα σεβαστοί. Συνεπώς λοιπόν το μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε είναι ότι η εθελοντική φύση της ε, ρύθμισης ε, δεν έχει αποδώσει. Είμαι 43 σήμερα και θυμάμαι όταν ήμουν νέα 16 ετών και προσπαθούσα να μάθω από πού προέρχονται τα ρούχα μου. Δεν είναι λοιπόν σωστό ε, να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε με τις εθελοντικές δραστηριότητες τώρα, λες και δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Νομίζω ότι για 30 χρόνια βλέπουμε ότι πάρα πολλές ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πιέζουν, αλλά δυστυχώς όμως ε, η ένδυση αντιπροσωπεύει, θα έλεγα, ένα να ελέγχουμε την παραγωγή ρούχων ακόμα και για νέα παιδιά που δεν έχουν πολλά χρήματα στη διάθεσή τους. I agree, I Συμφωνώ λοιπόν Πρόεδρε ότι υπάρχει ένα στενό σύνδεσμος επίσης ανάμεσα στην ανάπτυξη και την μετανάστευση. Αλλά δεν ήσασταν ξεκάθαρο στην απάντησή σας όταν είπατε ότι πράγματι βλέπουμε να υπάρχει μια κάποια χρηματοδότηση η οποία να πηγαίνει από την κανονική ανάπτυξη ε, στοχευμένη στην ε, μετανάστευση και αναφερθήκατε και στις συνοριακούς ελέγχους. Αλλά όπως είπατε αυτό δεν, οδηγεί, δεν πρέπει να οδηγήσει στη μείωση των ποσών για την εκρίζωση της φτώχειας. Αν πάρουμε λοιπόν χρήματα από την ανάπτυξη όπως γίνεται για να τα βάλουμε στη μετανάστευση και σε τομείς όπως η προστασία των σύνορων όπως είπατε, πώς αυτό δεν θα μειώσει τα, τις πιστώσεις ε, για την φτώχεια. Άλλοι τρει έχουν ζητήσει το λόγο. Σλάιν. Ευχαριστώ Επίτροπε για την παρουσία σας. Θα συμφωνήσω με την τελευταία ερώτηση της συναδέλφου Αργεντίνη. Πρώτον, θα ήθελα να πω ότι με χαρά σας άκουσα να αναφέρεστε στην πρωτοβουλία Collect More Spend Better Νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο εγώ ξέρετε ότι επιμένω πάρα πολύ, ιδιαίτερα στον τομέα της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες να το καταπολεμήσουν έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η πρακτική ικανότητα των χώρων αυτών. Ήδη εγκρίναμε για το θέμα αυτό μια έκθεση το 2015. Εσείς τι θεωρείτε, θεωρείτε ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές επηρεάζουν γενικά, έχουν συνέπειες για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μήπως εδώ υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης της συνοχικότητας των πολιτικών. Τον επόμενο χρόνο θα γίνει μια άλλη συζήτηση από ό,τι φαίνεται για το θέμα της μετατροπής της Επιτροπής Φορολογίας των Ηνωμένων Εθνών σε ένα πραγματικά γνήσιο διακυβερνητικό σώμα, έτσι ώστε και οι αναπτυσσόμενες χώρες να είναι στο ίδιο επίπεδο με τις αναπτυγμένες χώρες. Εσείς πριν την Άντις μας υπόσχεστε ότι δεν θα παρεμποδίσετε αυτό το πρώτο σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και έχουν πει κάτι ιδιαίτερα οι Σαρτζεντίνοι πει σημαντικό για την συνένεση ε, και τον σύνδεσμο ανάμεσα στη μετανάστευση και την ανάπτυξη. Θα ήθελα να σας ζητήσω να καταπολεμήσετε αυτή την τάση την οποία όλοι βλέπουμε και οι συνάδελφοι που ασχολούνται για τη μεταρρύθμιση στον τομέα του ασύλου, έτσι ώστε να υπάρξουν ισχυρές αιρεσιμότητες για τη βοήθεια, γιατί αυτό θέτει σε κίνδυνο τους στόχους που έχουμε για την ανάπτυξη ιδιαίτερα σε ένα διεθνές επίπεδο όπου πραγματικά τα SDGs κινδυνεύουν να μείνουν χαρτί άγραφο. Ε, πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να διατηρήσουμε τον ηγετικό μας ρόλο. Και δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται οι σχέσεις με τρίτες χώρες. Είδαμε τι έγινε βέβαια στην υπογραφή της συμφωνίας με κάποιες χώρες της Αφρικής για τη μετανάστευση και ιδιαίτερα να ευνοήσουμε τις χώρες οι οποίες είναι στον δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ξεχάσουμε τις προηγούμενες. Λέτε ότι το να, ξα... να ξοδεύουμε χρήματα στη μετανάστευση δεν σημαίνει ότι θα μειωθούν τα χρήματα για την ανάπτυξη. Πρέπει να το δούμε αυτό. Το Κοινοβούλιο αυτό θα πρέπει να έχει περισσότερε δυνατότητε ελέγχου έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι κάνουν όλα αυτά τα νέα χρηματοδοτικά μέσα και να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία, να δούμε τη λειτουργία του και να δούμε αν είναι συμβατά με το 208 του SDG. Η Επιτροπή μα έχει δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο μια συγκεκριμένη ομάδα εργασίας με στόχο να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ ε, και έχουμε άλλους δύο μιλητές. Μωρίς Πόγκο, πρώτος αντιπρόεδρος και μετά ο κύριος Κέγγε. Πρώτο ο κύριος Πόγκο Η κυρία Κέγγε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ μαζί μας. Θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα που πολύ με ασχολεί ε, σχετικά με το τελευταίο φόρουμ που έγινε στη Ρούμπα πέρυσι τον ε, ε, Φεβρουάριο. Το PTOM αναφέρε μια νέα εταιρική σχέση, σύγχρονη και στρατηγική με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, ήθελα να μάθω αν η Κομισιόν ε, έχει ε, ε, ασχοληθεί με το PTOM, δηλαδή τα υπερπόντια εδάφη και διαμερίσματα, ειδικά τώρα με το Brexit που υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο να προτείνει ένα νέο μηχανισμό που είναι ειδικό για τις υπερπόντες αυτές ε, περιοχές που θα βασίζεται σε ένα μηχανισμό όπως αυτόν που έχουμε για τη Γρινλανδία αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Σεσίλ Κέγκε, τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ Λίντα, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και για όλα όσα μας είπατε. Θα ήθελα να τονίσω δύο θέματα που σχετίζονται με την καλή διακυβέρνηση αλλά και με τη δημοκρατία. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με τους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Πόσο σημαντική είναι για σας και ποιες είναι οι πολιτικές που τους υποστηρίζουν. Τι θέλω να πω. Σχετίζονται άμεσα με τη δημοκρατία. Μια δημοκρατική χώρα πρέπει να είναι μια χώρα με ισχυρούς θεσμούς που θα μπορούν να αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε αλλαγή. Αυτό είναι δύσκολο σε πολλές χώρες. Έχουμε δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις αποστολές παρακολούθησης εκλογικών διαδικασιών ότι σε πολλές χώρες που βγαίνουν από σειράξεις όπως η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή η Μπουρκίνα Φάτσοσο η δημοκρατία ε, πηγαίνει αργά και είναι ακόμα σε δύσκολη θέση, θα λέγαμε. Το κοινοβούλιο, το κράτος ε, πρέπει να υφίστανται για να έχουμε έναν συνομιλητή. Η κυρία Σαρτζεντίνη ανέφερε ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με εμάς και με την διαφάνεια σε επίπεδο ηθικής. Υπάρχουν πολλές χώρες ε, ε, που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μιλάω, ας πούμε, για τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές ε, όπου υπάρχουν σειράξεις. Στην Δημοκρατία του Κονγκό πρόσφατα βρέθηκαν κάποιοι μαζικοί τάφοι. Τα τελευταία νέα που είχαμε ε, είναι ότι αυτή η τάφη ήταν σε περιοχές όπου έγιναν σφαγές ε, γιατί υπήρχαν και πάλι ε, ορυκτά. Άρα θα ήθελα να ξέρω οι μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε, πόσο σημαντικές είναι, ποια είναι η διαφορά που θα κάνουν. Αυτές οι μαζικές ε, δολοφονίες απλώς κρύβονται κάτω από το χαλί γιατί υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Πώς επηρεάζει αυτό λοιπόν τις κυβερνήσεις αλλά και τα, τα κινήματα. Ευχαριστώ. Και εγώ μια ερώτηση για τα φορολογικά. Ένα θέμα που έθεσαν πολλοί συνάδελφοι. Ο Θάμπο Μπέκη πέρυσι ήρθε στην Επιτροπή μας και μίλησε για την εργασία της Αφρικανικής Ένωσης όσον αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής. Είπατε ότι θα συνεργαστούμε και με άλλους για να έχουμε πρόοδο σε αυτό τον τομέα. Πολλά έχουν συμβεί από τότε που ήρθε σε πολλούς τομείς, αλλά ελπίζω ότι εντάξει, ε, αν ε, ε, πήγαμε στην Αντίς και υπογράψαμε την συμφωνία, αν δεν αντιμετωπίσουμε όμως αυτό το θέμα, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε από την Κομισιόν μια πρωτοβουλία για να διασφαλίσουμε ότι η Αντίς θα συμβεί τελικά, θα υπάρξει ε, πρόοδος. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Υπήρξε μια ερώτηση σχετικά με το πώς η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Πολιτική θα έχει επιπτώσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους και τις γυναίκες. Αυτό ήταν, είναι και θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των αναπτυξιακών μας στόχων είναι κομμάτι των προηγούμενων δραστηριοτήτων μας, αλλά και της νέας Ευρωπαϊκής Συμφωνίας και Συνένεσης για την Ανάπτυξη. Φέτος ε, οριστικοποιείται η ενδιάμεση αξιολόγηση το εισπροόδου που έχει γίνει. Ο σκοπός είναι να γίνει καλύτερη δρομολόγηση των προγραμμάτων έτσι ώστε να επιτύχουμε κάποιους από τους σημαντικούς αναπτυξιακούς στόχους που προκύπτουν από αυτή την συμφωνία, τη συνένεση για την ανάπτυξη. Αυτοί οι στόχοι θα έχουν ε, καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο δημιουργίας θέσεων εργασίας, ανάπτυξης, ενδυνάμωσης των γυναικών, ισότητας των φύλων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ε, ε, δράσεις για το κλίμα, συμπερίληψης του ιδιωτικού τομέα στις εταιρικέ σχέσεις. Όλοι αυτοί οι στόχοι πρέπει να μεταφραστούν σε δράσεις αναπτυξιακές από τα κράτη-μέλη και από την Επιτροπή. Έτσι λοιπόν θα γίνουν πράξη ε, εάν ανακατευθύνουμε τα κονδύλια στα εφιστάμενα ε, προγράμματα σε επίπεδο χώρας, ε, περιοχής για να έχουμε αποτελέσματα για το πλαίσιο μετά το κοτονού. Να επαναλάβω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι να εξετάσουμε την πιθανότητα τα κράτη-μέλη κυρίως γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς θα είναι η κατάσταση μετά το κοτονού, ποιο θα είναι το πλαίσιο. Όμως η Κομισιόν θα ήθελε η συζήτηση για αυτό το θέμα να κατευθυνθεί βάσει του δεσμευτικού νομικού πλαισίου της μελλοντικής ε, συμφωνίας που θα ενισχύσει όλες τις πτυχές της πολιτικής εταιρικής σχέσης, της σχέσεις ε, για την οικονομία και τον εμπόριο με όλες τις χώρες ΑΚΕ. Και μετά θέλουμε την ανάπτυξη τρίων συγκεκριμένων περιφερειακών πυλώνων με συγκεκριμένα ή λιγότερα, λιγότερο συγκεκριμένα ε, παραδείγματα για ειδικέ περιοχές της Αφρικής, του Ειρηνικού και της Καραϊβικής μέχρι το φθινόπωρο. Το αργότερο μέχρι τον Νοέμβρη θα μπορούμε να παρουσιάσουμε στο Συμβούλιο τις προτάσεις για τη διαπραγματευτική εντολή, δηλαδή τις οδηγίες διαπραγμάτευσης, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ε, για το πλαίσιο μετά το Κοτονού ε, μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι. Ο μηχανισμός τώρα που συμβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη. Η συνομοθετική διαδικασία έχει ήδη εκκινήσει. Το βέλτιστο σενάριο λέει ότι δεν θα τελειώσουμε πριν τον σεπτεμβριο οκτωβριο Φέτος το φθινόπωρο δηλαδή για τα ορυκτά που προέρχονται από ζώνες σειράξεων και τα συνοδευτικά μέτρα. Η εργασία ταυτοποίησης των μέτρων αυτών στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, για να υποστηρίξουμε τον κανονισμό για τα ορυκτά αυτά έχει ξεκινήσει, έχει αναπτυχθεί και συνταχθεί ένα νέο πρόγραμμα ανάπτυξης 5 εκατομμύρια ευρώ και συντονίζεται με τους διάφορους δωρητές και εταίρους, μεταξύ αυτών ε, την κοινωνία των πολιτών και τους ιδιώτες, τον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε για την βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων στις περιοχές ε, μετάλλευσης. Αντιμετωπίζουμε θέματα όπως η αναγκαστική εργασία, η παιδική εργασία, πολλά μέτρα συνοδευτικά που de facto θα, κάνουν, θα καταστήσουν δυνατή την ε, αναγνώριση της προέλευσης αυτών των ορυκτών έτσι ώστε να υπάρχει δέος επιμέλεια που ζητούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. 21 Ιανουαρίου είναι η ημερομηνία. Για την πρωτοβουλία σχετικά με την ένδυση και τα μέτρα Γνωρίζω πλήρως το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα, 27 Απριλίου. Ξέρω πολύ καλά τι λέει το Κοινοβούλιο. Απλώς πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει μια γρήγορη και εύκολη λύση για τις μεγάλες προκλήσεις του τομέα της ένδυσης. Πρέπει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Έχουμε παραδείγματα όπως το σύμφωνο του Μπαγκλατές, το πρόγραμμα καλύτερης εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με όλους αυτούς τους παράγοντες σε θελοντική βάση. Όλα αυτά φυσικά ε, θα μπορέσουν να φέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, ουσιαστικά αποτελέσματα. Αυτή είναι και η θέση μας. Λέμε λοιπόν απλώς ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο να βρούμε ποια θα είναι τα βέλτιστα αποτελέσματα βάσει της τρέχουσας διαδικασίας και των μηχανισμών που έχουμε στη διάθεσή μας ήδη. Ποιες είναι λοιπόν τι θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει εν το χρόνο να δούμε τα αποτελέσματα και με νομικά δεσμευτικούς ε, τρόπους να δώσουμε τη δυνατότητα για εθελοντική δράση. Τώρα, για το θέμα το κατά πόσο τα κονδύλια για τη μετανάστευση μειώνουν ή συρρυκνώνουν τα αναπτυξιακά κονδύλια για την εξάλληψη της φτώχειας, θα έλεγα... Θα έλεγα ότι η εξάλληψη της φτώχειας δεν θα γίνει μόνο με την επένδυσή μας σε παραδοσιακές, κλασικές, ατομικές ε, πολιτικές, αλλά με την ενίσχυση κρατικών θεσμών, με την επένδυση στην καταπολέμηση του εμπορίου ανθρωπίνων όντων, του σωματεμπορίου, με την επένδυση στη διαχείριση των συνόρων, επίσης συμβάλλουμε στην, στην εξάλληψη της φτώχειας. Με έμεσο τρόπο. Και δεν εξομοιώνεται η η εξάλληψη της φτώχειας μόνο με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ή την Επιτροπή ΔΑΚ. Αυτή είναι η κοινή αντίληψη περί και νέα αντιληψη βιώσιμης ανάπτυξης και η νέα προσέγγιση, μια πιο ε, διευρυμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη. Και μάλιστα τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε δείχνουν ότι δεν μειώνουμε την επίσημη αναπτυξιακή μας βοήθεια λόγω της χρηματοδότησης ε, το, της διαχείρισης των συνόρων που ούτως ή άλλως είναι περιορισμένη. Ε, από τα στοιχεία του 2016 για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια βλέπουμε ότι είχαμε το υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης και είχαμε πάνω από 75 δισεκατομμύρια ευρώ επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Περίπου το 60% της παγκόσμιας επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας προέρχεται από την ε, Ευρώπη. Οπότε ε, ο συνδυασμός της ανάπτυξης με τη μετανάστευση και την ασφάλεια δεν σημαίνει ότι θα συρρυκνώσουμε ή θα περικόψουμε τα κονδύλια για την ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά τα υπερπόντια δάφη και διαμερίσματα, Θα θέλαμε να διατηρήσουμε το ισχύον νομικό πλαίσιο, την απόφαση δηλαδή για τα υπερπόντια αυτά εδάφη και διαμερίσματα, μέχρι το τέλος της, του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και τότε θα είναι έτοιμο και το Κοινοβούλιο για να συζητήσουμε από κοινού το πιθανό νέο πλαίσιο για τα υπερπόντια εδάφη και διαμερίσματα εν ώψη του επόμενου πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου και μετά το 2020 δηλαδή. Προς το παρόν όμως διατηρούμε τους ισχύοντες μηχανισμούς και τα επιστάμενα μέσα σε ό,τι αφορά τη συνδρομή μας στην ανάπτυξη των υπερπόντιων εδαφών και διαμερισμάτων. Σε ό,τι αφορά τη φοροδιαφυγή, σίγουρα είναι πολύ σημαντική η καταπολέμησή της και στη συνένεσή μας για την ανάπτυξη, αλλά και σε όλες τις αναπτυξιακές μας δράσεις. Είμαστε έτοιμοι για συζήτηση με το Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη, τους ενδιαφερόμενους, για το πώς θα μεταφέρουμε τις αναπτυξιακές μας αρχές και αποφάσεις από την αναπτυξιακή μας πολιτική, πώς θα τις ε, μεταφέρουμε σε έμπρακτες ε, δράσεις, σε σχέδια δράσης πώς αποφάσει θα τι ε, εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα προκειμένου να καταπολεμήσουμε και τα φόρα διαφυγή στα πλαίσια των αναπτυξιακών μας στόχων. Σας ευχαριστώ Επίτροπε. Θα συνεχίσουμε το διάλογο μαζί σα. δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνουμε. Θα μπορέσουμε να δούμε ακριβώς τι θα γίνει με την ατζέντα post-Κοτονού για το μετά το Κοτονού το προσωπικό σας επεξεργάζεται το έγγραφο ε, με συγκεκριμένο τρόπο τι σημαίνει να καταλάβουμε γιατί υπάρχουν πολλές προσδοκίες για το τι πρέπει να γίνει γύρω από το θέμα αυτό της ε, αλυσίδας αξιών προσφοράς αναφερθήκατε ε, στα θετικά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο χρόνο και θα θέλαμε περισσότερα στοιχεία. Σας ευχαριστώ Επίτροπε. Σε ένα λεπτό θα περάσουμε στην υποδοχή του Επιτρόπου Στυλιανίδη. Περνάμε στο δεύτερο τμήμα της απογευματινής μας συζήτησης που προβλέπει τη σημαντική ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Στυλιανίδη στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου. Είπαμε ότι θέλουμε να εξετάσουμε το πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2018, ώστε να μπορέσουμε και εμεί να συμβάλλουμε με τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις προτάσεις μας προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα αξιόλογο πρόγραμμα εργασιών για το 2018 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλώς ήρθατε, είστε φίλος Επιτροπής, έχουμε στενή συνεργασία. και Ξέρω ότι αντιμετωπίζετε μια πολύ δυσχερή κατάσταση σε πολλές χώρες ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και θέλουμε να ακούσουμε περισσότερα για το έργο σας. Ξέρουμε ότι θέλετε να αναπτύξετε την αθεκτικότητα του συστήματος και συνεργάζεστε με τον Επιτροπό Μίμητσα για το δεσμό της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας με την ανθεκτικότητα και έχετε πολύ αξιόλογο έργο για τα προσφυγόπουλα. Αυτά έχετε το λόγο και μετά θα ακούσουμε τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ Λίντα. Αγαπητοί... Σας ευχαριστώ συναδέλφοι για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ίσως να γνωρίζετε ότι ήδη έχουμε ολοκληρώσει μαζί δυόμιση χρόνια, έχουμε διανύσει μαζί δυόμιση χρόνια. Σας είμαι ευγνώμων λοιπόν, επιδείξατε εξαιρετικό πνεύμα συνεργασίας και σας ευχαριστώ και για την ειλικρινέστατη φιλία σας. Όπως ε, έχω πάντα πει, ε, στην Επιτροπή σας ε, νιώθω σαν το σπίτι μου. Ταυτόχρονα, Είμαι υπερήφανος θα έλεγα γιατί η προσπάθεια που κάνουμε δείχνει να εκτιμάται δεόντως από τους ε, συμπολίτες μας που ενδιαφέρονται για τα θέματα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ε, ε, recent that we just published. This is good news. We need to Λοιπόν, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τα ευρήματα που μας λέγουν πώς είναι ικανοποιημένοι, να τα γνωστοποιήσουμε και να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από το σοβούν πολιτικό κλίμα, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες επαφές. Δυστυχώς όμως οι ανθρωπιστικές κρίσεις συνεχίζουν να κυριαρχούν στα εκατομμύρια των πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να θίξω τρία θέματα. Πρώτον, να πω τι κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή. Δεύτερον, να προσπαθήσω να αναφερθώ στα βήματα προόδου τα οποία έχουμε επιτελέσει και τέλος να μιλήσω για τους τομείς της πολιτικής τους οποίους συγκεντρώνουμε την προσοχή μας. Μία από τις βασικές προτεραιότητες ε, είναι να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τις ανθρωπιστικές συνέπειες της προσφυγικής κρίσης και σε τρίτες χώρες αλλά και στο εσωτερικό ε, των συνόρων μας. Αυτή είναι και δική σας προτεραιότητα. Μέσω του, ακριβώς με το μέσο αυτό της κατεπίγουσας στήριξης ε, προσπαθούμε να βοηθήσουμε και βοηθάμε 62.000 πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα. Καταθέσαμε και την ετήσια εκθεσή μας, η οποία είναι στην διάθεσή σας. Μέχρι τώρα ε, δώσαμε καταφύγιο και ε, τρόφιμα σε πάνω από 35.000 πρόσφυγες. Τους δώσαμε επίσης προπληρωμένες τηλεφωνικές κάρτες για να καλύψουν τις ανάγκες τους οι ίδιοι με αξιοπρέπεια μόνοι τους. Υποστηρίξαμε τα συστήματα εκπαίδευσής τους, δημιουργήσαμε 450 χώρους επίσης για ασυνόδευτους ανήλικους. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι η κατάσταση στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην υπηρετική χώρα, ε, ότι έχει βελτιωθεί, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό αλλά παραμένουν πάρα πολλές δυσκολίες και μένει να γίνουν πολύ περισσότερα. Με έναν προϋπολογισμό 250 εκατομμυρίων ευρώ φέτος θα πρέπει να μετακινήσουμε ε, πρόσφυγες από ε, τις σκηνές σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες έμου ε, του ιδίου και των υπηρεσιών μου και να προσπαθήσουμε επίσης να περάσουμε από τη λογική του εξωτερικού υπεργολάβου catering σε μετρητά για αγορά τροφίμων. Έτσι θα γίνουν όλα πιο αποτελεσματικά. Η υποστήριξη των προσφύγων είναι βασική μας προτεραιότητα επίσης και στην Τουρκία. Όπως είπα, το μέσο αυτό Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι ο πιο σημαντικός πυλώνας στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε για να αντιμετωπίσουμε με την κρίση των προσφύγων. Άνω των 2,9 δις από τα τρία που είχαν ε, υπολογιστεί για το 16 και 17 έχουν ήδη κινητοποιηθεί και όλα αυτά μέσα μόνο σε ένα χρόνο. 790 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη δαπανηθεί αυτό έγινε σε ταχύτατους χρόνους, με διάφανο τρόπο, με ελεγχόμενο τρόπο. Ε, βασικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων για τους πρόσφυγες. Ε, συζητήσαμε ήδη το ESSM, το πρόγραμμα του κοινωνικού ε, έκτακτου δικτύου, το οποίο είναι στην καρδιά της προσπάθειας μας στην Τουρκία το ταμείο αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει χρηματοδοτήσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των ανθρωπιστικών. 348 εκατομμύρια ευρώ ο αρχικός προϋπολογισμός και θα φτάσει πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες μέχρι το καλοκαίρι. Αγαπητοί συνάδελφοι, να μου επιτρέψετε τώρα να έλθω στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Η κρίση στη Μέση Ανατολή πράγματι δεν μας κάνει να είμαστε δυστυχώς πολύ αισιόδοξοι. Η τραγική κατάσταση στην Συρία είναι δυστυχώς πέραν κάθε ελέγχου και στο Χαλέπι και σε άλλες περιοχές Άνω των 13 εκατομμυρίων σύρων έχουν ανάγκη εκτακτής ανθρωπιστικής βοήθειας, μεταξύ των οποίων τα 6 εκατομμύρια είναι εκτοπισμένοι εσωτερικά. κάθε ε, θα έλεγα περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μία περισσότερο από όσο πρέπει ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες ε, για τους πρόσφυγες όπως επιβεβαιώθηκε ε, και στην διάσκεψη που έγινε εδώ στις Βρυξέλλες τον μήνα Απρίλιο. Αυτός είναι βασικός μας στόχος. Εγώ επανειλημμένα έχω πει ότι θα πρέπει να υπάρξει για τέτοιου είδους εγκλήματα ανάληψη ευθύνης με βάση τους ισχύοντες διεθνείς νόμους και τις ε, αποφάσεις του Συμβουλίου Αυστραλίας. Στα πλαίσια της νέας στρατηγικής μας για τη Συρία έχουμε επαναλάβει την θέση μας. Δεν θα υπάρξει στήριξη οικονομική για την ανοικοδόμηση αν δεν έχει διασφαλιστεί η ειρηνική και δίκαιη μετάβαση από τους ίδιους τους Σύρους. Στο Ιράκ, όπως γνωρίζετε, επισκέφτηκα την χώρα αυτή τέσσερις φορές. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες σύρους αμάχους γύρω από την πόλη της Μοσούλης, ιδιαίτερα την Ανατολική Μοσούλη. Καταφέραμε να μείνουν στις κατοικίες τους οι άνθρωποι αυτοί χάρη στον θετικό τρόπο με τον οποίο οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ ε, ε, διεξήγαγαν τις πολεμικές τους επιχειρήσεις. Πήγα εκεί και διαπίστωσα τον θετικό ρόλο τον οποίο έχουν παίξει ε, οι αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας έτσι ώστε να επιβάλλουν ουσιαστικά στις δυνάμεις ασφαλείας να συμπεριφερθούν σύμφωνα και συμβατά με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Για μένα ήταν μια έκπληξη αυτό, αλλά ήταν ταυτόχρονα και ένα ιδιαίτερα θετικό μήνυμα. Οι εταίροι μας λοιπόν επί τόπου προσπάθησαν να πείσουν τις δυνάμεις ασφαλείας και βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι πλέον απτά. Στην δυτική Μοσούλ όπου εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι 450.000 άμαχοι, τον ΤΑΕΣ ε, χρησιμοποιεί πάντα τους αμάχους ως πως ανθρώπινες ασπίδες και δυστυχώς ε, ε, αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, πολλοί προσπαθούν να διαφύγουν με πολλά θύματα και απαιτείται προσπάθεια από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ για τον σεβασμό των αμάχων και τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Παραλλήλα, σε σχέση με το IHL, ε, ο συντονισμός ανάμεσα στις πολιτικές υπηρεσίες και τις στρατιωτικές δυνάμεις είναι απαραίτητος. Uh, Σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο λοιπόν. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε με σωτήριο τρόπο θα έλεγα τους παγιδευμένους ε, ε, αμαχούς. Από την αρχή της κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους βασικούς δωρητές 159 εκατομμύρια δώσαμε μόνον πέρυσι. Ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει ιδιαίτερα και στην κατεπίγουσα ιατρική ε, βοήθεια. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ κοντά στην πόλη της Μοσούλης ένα κινητό νοσοκομείο και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος ε, όπως και όλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα σε αυτήν την ανάληψη ευθύνη στον ιατρικό τομέα. Έτσι λοιπόν η βοήθεια αυτή είναι απαραίτητη έτσι ώστε να σωθούν πλέον ζωές. Ταυτόχρονα ε, επιτρέπει στο μέλλον να υπάρξει διαρκή ειρήνη και συμφιλίωση στην χώρα. Αναφέρθηκα στο ρόλο της ανθρωπιστικής βοήθειας σε σχέση με την διαδικασία συμφιλίωσης Πέρα από το Ιράκ αυτό που μας ανησυχεί είναι οι σειράξεις στην Ιεμένη με τρομερές ανθρώπινες και οικονομικές συνέπειες. Ο πόλεμος δυστυχώς έχει οδηγήσει στην μεγαλύτερη κατεπίγουσα κατάσταση στον τομέα της έλλειψης τροφίμων. Αυτή η έλλειψη τροφίμων επηρεάζει άνω των 17 εκατομμυρίων πολιτών και ε, ε, τα 7 εκατομμύρια βρίσκονται σε κατάσταση τροφοδοτικής ανασφάλεια ανασφάλειας και έχουν ανάγκη από άμεση βοήθεια. Η διάσκεψη για την Ιεμένη στη Γενέβη την προηγούμενη εβδομάδα, στην οποία ήμουν παρόν, μπόρεσα να διαπιστώσω ότι υπάρχει ε, κάποια, κάποια ελπίδα εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε τους Ιεμενίτες. Όλες οι αντιπροσωπείες που ήσαν παρούσες στην Γενέβη φτάσαμε το ένα δις, η υπόσχεση ένα δις για τη στήριξη του πληθυσμού α, κατά τη διάρκεια του 2017. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή α, προτείνει και υπόσχεται 116 εκατομμύρια και το 50% του συνόλου των υποσχέσεων προήλθε από το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μεμονωμένα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τώρα να ξεπεράσουμε απλά τις δηλώσεις, να σεβαστούμε τις υποσχέσεις αυτές, έτσι ώστε να μετριάσουμε τον λοιμό ο οποίος πέφτει, έρχεται μάλλον, και πέρα από την Ιεμένη η Σομαλία, το Νότιο Σουδάν και η Νιγηρία αντιμετωπίζουν και αυτές προβλήματα σοβαρών συνθήκων έλλειψης τροφίμων. Η κρίση αυτή είναι δυστυχώς ανθρωπογενής, απολύτως ανθρωπογενής. Άνω των 20 εκατομμυρίων πολιτών στις τέσσερις αυτές χώρες αντιμετωπίζουν το φάσμα της πείνας είναι η μεγαλύτερη διατροφική κρίση από την δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών μέχρι σήμερα. Η πρόσβαση στις περιοχές αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολη λόγω των σειράξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Από τις πρώτες προειδοποιήσεις στον βόρειο-ανατολική Νιγηρία στο τέλος του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιταχύνει την ροή πιστώσεων και έχει κάνει διάφορες δράσεις, έχει αναλάβει διάφορες δράσεις συνειδητοποίησης του προβλήματος. Τον προηγούμενο Φεβρουάριο πήρα μέρος στην συνάντηση στο Όσλο για την κρίση γύρω από την λίμνη Τσάδ. Σαν Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε υποσχεθεί και εκεί είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής 105 εκατομμύρια ευρώ. Τον προηγούμενο μήνα εμείς ανεβήκαμε στην κλίμακα προειδοποίησης αν θέλετε με ένα επιπλέον ποσό 165 εκατομμυρίων ευρώ βοηθώντας την Σομαλία και τον Νότιο Σουδάν που έχουν μεγάλες ανάγκες σε επίπεδο πείνας και θα πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα προσπάθειες για να υποστηριχθεί η επιβίωση των πληθυσμών και η γρήγορη ανάκαμψη προωθώντας την ανθεκτικότητα του ε, πληθυσμού που φύγεται από τις συνθήκες αυτές. Ο συνδυασμός της διασφάλισης των ε, τροφίμων ε, και των δυνατοτήτων επιβίωσης, η συνεργασία μας με τον Διεθνή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων συνεχίζεται και επαναλαμβάνω ότι η βασική μας προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση του λοιμού, χωρίς να ξεχνάμε άλλες κρίσεις που φύγουν την ζωή χιλιάδων πολιτών στο Μαλί ή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Πιο κοντά σε μας, πιο κοντά στην Ευρώπη, βοηθάμε επίσης και τον πληθυσμό, ο οποίος θίγεται από τη σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία η ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία είναι μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ επισκέφθηκα τη χώρα αυτή τον προηγούμενο Φλεβάρι και επιβεβαίωσα την αλληλεγγύη μας με τα πιο ευάλωτα κομμάτια του πληθυσμού. Δεν μπορούμε εμείς να αφήσουμε την Ουκρανία να μετατραπεί σε ε, χώρα χαμένη και ξεχασμένη. Είμαστε από τους βασικούς δωρητές στην Ιεμένη και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτούς που υποφέρουν από τη σύγκρουση αυτή όσο και να χρειαστεί. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, το πρόβλημα στο Αφγανιστάν δυστυχώς χειροτερεύει. Υπάρχουν ε, πολλά θύματα ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό και τους εργαζομένους της ΜΚΟ. Αυξάνεται ο αριθμός των εκτοπιστέντων και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να ανησυχούμε. Μέσω της συνεργασίας ε, με τον συνάδελφο επίτροπο Μίμητσα, ε, εμείς συνδυάζουμε τις προσπάθειες των υπηρεσιών μας όπως επίσης και με την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών και το IOM, έτσι ώστε την Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις δύσκολες συνθήκες. Πριν από μερικούς μήνες επισκέφτηκα και το Ιράν. Είδα με θετικό τρόπο το πώς αντιμεταπίζουν το 3 εκατομμύρια Αυγανών προσφύγων που έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και σε ε, ιατρική φροντίδα. Ήταν ένα πολύ θετικό μήνυμα αυτό που πήρα από το Ιράν. Θα ήθελα η κατάσταση αυτή να συνεχιστεί λοιπόν και μετά από τις αλλαγές σε πολιτικό επίπεδο και τις αλλαγές ε, ε, στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και την αντίδραση της κυβέρνησης των ΗΠΑ στη λεγόμενη συμφωνία με το Ιράν. Παρακολουθώ επίσης πάρα πολύ προσεκτικά την ανθρωπιστική κατάσταση στην Μαρ. Χτες με τη Φεντερίκα Μογκερίνη συναντηθήκαμε με ε, τον ε, σύμβουλο της ε, Σούνκι την συνεχάριμεν για τις εξαιρετικές ε, προσπάθειες που έκανε για την ε, συνέχιση των δημοκρατικών διαδικασιών. Είναι πραγματικά ένας ήρωας ε, σε σχέση με τη δημοκρατική μετάβαση. Αλλά όμως εκφράσαμε σε βάθος την ανησυχία μας για την, για την κατάσταση που χειροτερεύει στις βόρειες πολιτείες της Μιανμάρ από το προηγούμενο φθινόπωρο και μετά. Να κάνω επίσης μια ανακοίνωση μετά από συμφωνία με τον σύμβουλο, τον επίσημο σύμβουλο της κυβέρνησης της Μιανμά. Θα επισκεφτώ τη Μιανμάρ την επόμενη εβδομάδα. Αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη ενός ε, Ευρωπαίου Επιτρόπου στην χώρα αυτή. Θα συναντηθώ με τις τοπικές επίσης αρχές και με τους υπουργούς και θα δούμε από κοντά τι μπορούμε να κάνουμε. Αποφάσισα να κάνω την επίσκεψη αυτή γιατί γι' αυτό υπάρχουμε και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ανθρωπιστικές μας αρχές είναι η μοναδική μας ε, οδηγή. Βοηθάμε αυτούς που το έχουν ανάγκη ανεξάρτητα ε, του θρησκευματό τους, ε, της ε, φυλής τους, της τοποθεσίας στην οποία ζουν. Είναι ηθικό μας καθήκον να το κάνουμε. Αγαπητοί φίλοι, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής δυστυχώς και αυτές αντιμετωπίζουν κρίσεις όπως και η Καραϊβική. Οι φυσικές καταστροφές τους πρώτες μήνες του 2017 δείχνουν πόσο εκτεθειμένη είναι η περιοχή αυτή σε φυσικές καταστροφές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη πρόσφατα αντιμετώπισε τις δασικές πυρκαγιές στη Χιλή, τις πλημμύρες στο Περού, όπως επίσης και τις κατολιστήσεις στην Κολομβία. Η απάντησή μας στην κρίση στη Λατινική Αμερική έχει αποδείξει για μια ακόμη φορά τον κρισιμότατο ρόλο του μηχανισμού πολιτικής άμυνας. Ταυτόχρονα, και θυμάμαι κυρία Μακάβαν την επίσκεψή μας πριν μερικά χρόνια, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον σημαντικό ρόλο του Κέντρου Συντονισμού Άμεσης Ανταπόκρισης στις Βρυξέλλες. Είναι ένα κρίσιμο μέσο το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά και στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Μας βοηθά το μέσο αυτό να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις κρίσεις και να σεβαστούμε και να σεβαστούμε τις προσδοκίες των συμπολιτών μας. Είχαμε πάει μαζί Λίντα, είδες πραγματικά τι σημαντική δουλειά κάνουμε από την πλευρά του ERCC. και η σημαντική αυτή δουλειά του Μηχανισμού Πολιτικής Άμυνας υπογραμμίστηκε και από το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο. Μέχρι το τέλος του Μαΐου θα λάβουμε κάποιες περαιτέρω εκτιμήσεις για τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας μέσω μιας συνεχιζόμενης εξωτερικής αξιολόγησης η οποία θα έρθει την κατάλληλη στιγμή. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα ταιριάξει με τις διαδικασίες τις οποίες ακολουθούμε για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου 2020-2027. Σε τρεις εβδομάδες θα μεταβώ στο Μεξικό για την πέμπτη παγκόσμια πλατφόρμα για την αποτροπή των ε, καταστροφών. Και νομίζω ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την όθηση που έχουμε πάρει για να προωθήσουμε και στην Ήπειρό μας αλλά και παγκοσμίω αυτή την πρωτοβουλία και θα είμαι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ενωσιακής Αντιπροσωπείας. Θα διδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στη διάσκεψη αυτή, συμμετέχοντας ε, σε όλες τις επιμέρους ομάδες και πάνελ και μάλιστα και ο Έρικε Γκερέρο Σαλόν που είναι μόνιμος συγκητής για την ανθρωπιστική βοήθεια δέχτηκε την πρόσκλησή μου και θα συμμετάσχει και αυτός στην ε, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μεταβεί στο Κανκούν. Αυτό είναι μια άλλη απόδειξη της ε, συνεχούς δέσμευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μείωση του κινδύνου από καταστροφές. Επιτρέψτε μου τώρα να σταθώ λίγο στις προτεραιότητες μας για το έγκυς μέλλον. Καταρχήν, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε εκπαίδευση στα παιδιά που έχουν πληγεί από την προσφυγική κρίση. Αυτό είναι προτεραιότητα, είναι σχεδόν ιδεολειψία μου. Ε, αυτή είναι προτεραιότητα και όπως ε, έχει δείξει και η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, 91% των Ευρωπαίων πολιτών στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν ε, ενδιαφέρει και τους πολίτες γιατί η παιδεία, ε, οι ανάγκες για την παιδεία είναι τεράστιες και δυστυχώς δεν έχουν τύχει τη δέσους προσοχής ούτε αποτελούν προτεραιότητα σε πολλές κρίσεις και πραγματικά ελπίζω και εύχομαι να αλλάξει αυτή η τάση. Και εμείς θα πρωταγωνιστήσουμε στην αλλαγή αυτών των τάσεων, ώστε να δοθεί δέουσα προτεραιότητα στην παιδεία και να ικανοποιηθούν οι τεράστιες ανάγκες που έχουμε στην παιδεία. Και με την δική σας ουσιαστική βοήθεια δαπανούμε πάνω από το 4% του προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας ε, το 2016 και φέτος ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο 6% της ανθρωπιστικής βοήθειας για, τη χορήγηση των για την χρηματοδότηση εκπαιδευτικών αναγκών. Και κυρίως επιτόπου βλέπουμε αλλαγέ με αυτή τη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού. Το βλέπω με τα μάτια μου σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, στην Τουρκία, με 34 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμά μας, το Μάρτιο εγκαινιάσαμε μαζί με τη UNICEF ε, πρόγραμμα που ε, βοηθά 230.000 προσφυγόπουλα για να μορφωθούν. Στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκή επικράτεια δηλαδή, διευκολύνουμε την μεταφορά 2.000 ε, παιδιών προσφυγόπουλων σε σχολεία και φυσικά στηρίζουμε και την επίσημη εκπαίδευση και τις σχετικές δραστηριότητες για 9.000 παιδιά. Έχουμε πολύ άριθμα παραδείγματα από το Ιράν μέχρι την Ιγυρία, αλλά και στη Μιαμάρ. Γι' αυτό θα επισκεφθώ και την επόμενη εβδομάδα ένα δικό μας πρόγραμμα στη Μιανμάρ που επικεντρώνεται στις έκτακτες ανάγκες στον τομέα της παιδείας. Αγαπητοί φίλοι, πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την άγωψα. Δύσκολος ο δρόμος μας, αλλά είναι καθήκον μας να το κάνουμε, γιατί ο αντίκτυπος ε, των, του, των ποσών αυτών είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι περιμέναμε, ο θετικός αντίκτυπος. Και φυσικά ε, δεύτερο θέμα, θα συνεχίσουμε σε όλες μας τις πολιτικές προσεγγίσεις που θα εδράζονται στην ανθεκτικότητα για να ενισχύσουμε καταρχήν τους δεσμούς μεταξύ αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Και είμαι βέβαιος ότι ο αγαπητός συνάδελφος Νέβεν Μίμητσα ήδη το ανέφερε, ήδη ανέφερε αυτό το στενό δεσμό, γιατί το συζητήσαμε εκτενώς και σε πολλές περιπτώσεις πώς να βελτιώσουμε ακριβώς αυτό το δεσμό, πώς να το κάνουμε πιο στενό, αυτό το δεσμό μεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας. 14 χώρες έχουν εντοπιστεί για πιλωτικά προγράμματα με αυτό το περιεχόμενο. Και στόχος μας είναι να, να διεξάγουμε μια κοινή ανάλυση των κινδύνων και των ευπαθειών, των τροτών σημείων, ώστε να καταλήξουμε στις βέλτιστες πρακτικές για να αναπτύξουμε και περαιτέρω εταιρικέ σχέσεις με βασικούς παγκόσμιους φορείς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και τα Ηνωμένα Έθνη. Για μένα είναι αρκετά σημαντικό και για τον Εύεν Μίμητσα το ίδιο να διαπιστώνουμε και στην πράξη και επιτόπου αυτό το στενό δεσμό ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας σε όλες τις πτυχές των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών μας δράσεων. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για τη συνεχή σας υποστήριξη στον προϋπολογισμό μας για την ανθρωπιστική βοήθεια φέτος το 2017 από έναν αρχικό προϋπολογισμό 936 εκατομμύριων ευρώ φτάσαμε στα 1,8 δις ήδη. Αισθητή αύξηση του προϋπολογισμού, χάρη και στη δική σας συνδρομή. Εν όλων αυτών λοιπόν, του χρόνου οι προβλέψεις ε, επαρκών επιπέδων ανθρωπιστικής ε, ενίσχυσης θα εξακολουθούν να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για συγκεκριμένο λόγο, αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να είναι πρωταγωνιστής και να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες με επαρκή προπολογισμό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση που μου απευθύνετε και για την προσοχή. Ακούσατε τις προπτικές μας, τις προκλήσεις μας, τα σχέδιά μας και όπως πάντα υπολογίζω γενικώ στην στήριξή σας, στη βοήθειά στη συνεργασία σας και περιμένω τις παρατηρήσεις σας, τις απορίες σας, αλλά και τις επικρίσεις σας, την κριτική σας. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Μας κάνατε μια ευρή επισκόπηση του έργου σας και χαίρομαι ιδιαίτερος που θα μεταβείτε στη Μιανμάρ, γιατί γνωρίζουμε ότι η Αν Σανξουκή που έχει βραβευτεί με το βραβείο Ζαχάροφ είναι μια προσωπικότητα που σεβόμαστε ιδιαίτερος και Ξέρουμε τι γίνεται με το, το λαό ε, Ροχάν, και θα πρέπει να, να αντιμετωπιστεί Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα στη Μιανμάρ. Και σήμερα συναντήθηκα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιεμένης, γιατί αναφερθήκατε στην Ιεμένη. Εκατομμύρια άνθρωποι τη στιγμή που μιλάμε χάνουν τη ζωή τους στην Ιεμένη. Και θα πρέπει να ανοίξουμε ανθρωπιστικούς διαδρόμους παρά τις τεράστιες πολιτικές δυσκολίες. Φαντάζομαι οι συνάδελφοι θα έχουν πληθώρα ερωτήσεων να σας υποβάλουν. Θα ξεκινήσουμε από τον μόνιμο εισηγητή μας για την ανθρωπιστική βοήθεια, τον Ερίκη Γκερέρο Σαλόμ και μετά Έγγελ Χόιμπουχ, Βέντα Χόιμπουχ, Χιμένες και Κέγγε. Αν θέλει και κάποιος άλλος να το δηλώσει, γιατί σε έξι ακριβώς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Eh, eh, Ευχαριστώ. Εδώ και πολλά χρόνια, πέντε αν δεν κάνω λάθος, ε, ήμουν ο συντονιστής της πολιτικής μου ομάδας για το ψήφισμα με θέμα το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, πρωτοστάτησε διαπραγματεύσεις με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Οπότε εκ γνωρίζω ότι δεν ε, ε, θα αφήσουμε να είναι, μικρό το, η παρά, δεν είναι μικρή παράγραφος για την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανθρωπιστική πολιτική. Τέτοιου είδους ε, ευκαιρίες όπως η σημερινή, ανταλλαγή απόψεων, είναι πολύ σημαντικές γιατί μία παράγραφό ενό ψηφίσματο που περιλαμβάνει και άλλε προτεραιότητε δεν είναι δυνατόν να εξαντλήσει το θέμα. Και είναι δύσκολο να προτάξουμε τι δικέ μα προτεραιότητες. Γι' αυτό και χαίρομαι για την ευκαιρία που σήμερα μα δίνεται να επεκταθούμε στα θέματα αυτά. Και επίση είναι ικανοποιητικά τα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου. Γνωρίζουμε ότι όταν ερωτούνται από το Ευρωβαρόμετρο παρά είναι γενναιόδορε απαντήσει τους, πολύ πιο γενναιόδοροι από ό,τι στην πραγματικότητα. Κανένα σε μια δημοσκόπηση δεν λέει με κατά τη ανθρωπιστική βοήθεια. Τα στοιχεία όμως παρόλα αυτά δείχνουν ε, με σαφήνεια ότι η αλληλεγγύη των Ευρωπαίων πολιτών είναι μεγαλύτερη και πιο σημαντική από την αλληλεγγύη των κυβερνήσεων των κρατών μέλων. Και αυτό το διαπιστώσαμε σε όλες τις κρίσεις. Και είναι θετικό να απευθύνουμε έκκληση άμεσα προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Ακόμη και αν τα πραγματικά ποσοστά είναι κάτω από το 80-90% που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις στο Ευρωβαρόμετρο. Ο Επίτροπος ε, μας ε, έκανε μια λεπτομεριακή επισκόπηση, ένα ταξίδι σε όλες αυτές τις κρίσεις που μαστίζουν τον πλανήτη μας και σχεδόν σε όλες αυτές τις κρίσεις ε, έδωσε το παρόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλίες, με ψηφίσματα, με υποβολή ερωτήσεων, με διεξαγωγή συζήτησης. Και σε όλες τις περιπτώσεις, νομίζω, στηρίξαμε το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα το έργο του Επιτρόπου. Και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αυτό να το υπογραμμίζουμε, γιατί πραγματικά έχουμε στενή συνεργασία σε ένα τομέα που απαιτεί συντονισμό και αμοιβαία υποστήριξη για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τις ανθρωπιστικές. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες του 2018, θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε την ε, συνένεση για την ανθρωπιστική βοήθεια με ένα νέο σχέδιο δράσης και ίσως αυτό θα ήταν ε, μία άλλη, ε, ένας άλλος τομέας που θα μπορούσε να μας απασχολήσει για το επόμενο έτος και να τον αναπτύξουμε. Ήδη έχουμε ζητήσει από τον Επίτροπο, το επαναλαμβάνω το αίτημα αυτό και επισήμω σήμερα, ε, κάποια στιγμή, μέσα στο 2017, να μας ετοιμάσετε μία αξιολόγηση ε, για να δούμε σε ποιο βαθμό τηρούνται οι δεσμεύσεις ε, που αναλύθησαν στην Κωνσταντινούπολη και από τα κράτη-μέλη ε, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαμορφώσουμε μία ιδέα για το ποια είναι η πρόοδος μας στα διάφορα θέματα και στους διάφορους τομείς για τους οποίους έχουμε αναλάβει δέσμευση στην Κωνσταντινούπολη. Και φυσικά θα συνεχίσετε να λαμβάνετε και τη δική μου προσωπική βοήθεια και συνδρομή, αλλά και την στήριξη της ομάδας μου, αλλά και άλλων πολιτικών ομάδων, τη βοήθειά μας ώστε ο προϋπολογισμός για την παιδεία και για τις έκτακτες ανάγκες στην παιδεία ε, δεν αυξηθεί, τουλάχιστον να διατηρηθεί στα φετινά επίπεδα. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω, αν κάποιος το ξεχάσει, 6% σημαίνει τριπλασιασμό του ποσοστού που είχαμε κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής θητείας. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε στο Ε, να το αναγνωρίσουμε γιατί οφείλεται μέσα στο έργο του Επιτρόπου αλλά και στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό ο τριπλασιασμός του ποσοστού στον προϋπολογισμό. Είπατε ότι σε περίπτωση που γίνονται επιθέσεις ε, σε ε, προσωπικό μοικιό ή σε εγκαταστάσεις ΜΚΙΟ θα πρέπει να προωθήσουμε μια πολιτική πρωτοβουλία για να επιληθεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Συμφωνώ. Είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο και επιπλέον πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να προτείνουμε από κοινού με τους ανθρωπιστικούς φορείς και τις οργανώσεις, ε, τις ανθρωπιστικές παγκοσμίω, μια στρατηγική για το σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του σεβασμού των αρχών της προστασίας του προσωπικού των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχειώδες καθήκον, ένα θεμελιώδες καθήκον που έχουμε απέναντι στις οργανώσεις αυτές. Θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, ξεχασμένες κρίσεις ή στις ε, κρίσεις που δεν βρίσκονται ε, στο επίκεντρο της προσοχής μας. Σήμερα είχα μία συνάντηση με εκπροσώπους του, διεθνούς, ε, του, του Δανέζικου και του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων και με την International Relief και μου ανάφεραν την περίπτωση του Ιράν και την περιοχή που επισκεφτήκατε. Μου εξήγησαν και οι εκπρόσωποι αυτών των οργανώσεων ότι 3,5 εκατομμύρια Αφγανοί είναι οι πρόσφυγες στο Ιράν και η βοήθεια που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή που λαμβάνουν η Τουρκία, ο Λίβανος ή η Ορδανία για αντίστοιχο πληθυσμό. Και το λέω όχι γιατί πρόκειται για το Ιράν, γιατί, αλλά γιατί υπάρχουν κρίσεις που για την κοινή γνώμη φαίνεται να μην υπάρχουν. Αλλά 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι Αυγανοί είναι διόλου μελιτέο. διόλου αριθμός. Επίσης θα πρέπει να στηρίξουμε την ανθρωπιστική μεταχείριση αυτών των προσφύγων. Κάτι τέτοιο θα συμβάλλει και στην πολιτική σταθερότητα του Ιράν που μας ενδιαφέρει και παγκοσμίω αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας στόχος πρώτης τάξης για την παγκόσμια ειρήνη. Οπότε θα πρέπει να δούμε σε τι βαθμό μπορούμε να αυξήσουμε την ενίσχυση προς το Ιράν για την ανθρωπιστική μεταχείριση των εκατομμύριων αυτών αυγανών προσφύγων. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τη Λατινική Αμερική, ξέρω ότι γίνεται ένα συντονισμό των εθνικών μέσων των κρατών μελών με τα ευρωπαϊκά μέσα, με τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρόσφατα ήσασταν στην Ισπανία και επισκεφθήκατε την στρατιωτική μονάδα έκτακτη ανάγκης που έστειλε πυροσβέστε στη Χιλή για τις προσπάθειες κατάσβευση ε, των πυρκαγιών. Ε, ένα ξεκάθαρο παράδειγμα συνεργασίας ε, εθνικών δράσεων με ευρωπαϊκές. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω κάτι που αξίζει επισήμασης. Το Είπατε και εσείς κύριε Επίτροπε ότι με προσκαλέσατε να λάβω μέρος στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Κανκούν για, την, για τον περιορισμό των, των, των κινδύνων καταστροφών. Αυτή όμως η πρόσκληση δεν έγινε προσωπικά σε μένα τον Ερίκε Γκερέρο, αλλά είναι μια πρόσκληση προς την Επιτροπή της ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης και μέσω του μόνιμου συγητή είναι μια ε, πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για συμμετοχή και συνεργασία σε προτεραιότητες τις οποίες εστερνιζόμαστε και να συμμετέχουμε σε δράσεις που μπορούμε, ε, με τις οποίες μπορούμε είτε να μετριάσουμε τα δεινά είτε να τα αποτρέψουμε σε ό,τι αφορά καταστροφές. Ε, και σας ευχαριστώ κύριε Επιτρόπε που με εμπλέξατε και μένα ε, και με προσκαλέσατε σε αυτή την εκδήλωση στο Κανκούν. Ευχαριστώ. Έχουμε αρκετού ομιλητέ. Δύο λεπτά παρακαλώ ο καθένα και περιοριστείτε ε, σε ερωτήσεις στο μέτρο του δυνατού. Ο Φράγκα Έγγελ είναι ο πρώτος ομιλητής. Ε, Ευχαριστώ, Λίντα. Α το κάνουμε όπω όταν είμαστε στην Ολομέλεια και να τελειώνουμε σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ, ε, κύριε Επίτροπε, για την αδιάκοπη παρουσία σας σε αυτό το Tour αυτή την πολύ σημαντική παρουσίαση για όλα τα θέματα και ειδικά σε επίπεδο περιεχομένου. Υπάρχουν θέματα που μπορούμε να ασχοληθούμε πιο επισταμένα. Ε, ας πούμε για την Τουρκία. Θυμάμαι όταν η Λίπε πήγε εκεί, μίλησε ε, για τους ε, ανθρωπιστικούς ακτιβιστές και για τους πρόσφυγες και μιλούσαμε εκεί για το πρόγραμμα διατροφής το οποίο ε, ήταν ε, μεγάλο, ήταν 300.000 ε, άνθρωποι εκεί και έλειπαν περίπου 3 εκατομμύρια γι' αυτό, όχι δις. Αν μπορούμε να κινητοποιήσουμε, ξέρω ότι υπάρχει αυτή η δήλωση, αλλά αν μπορούμε να κινητοποιήσουμε ένα ή δύο ή τρία δις για να βοηθήσουμε αυτούς τους πληθυσμούς ως Ένωση, θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε και τις εισφορές που πηγαίνουν στο παγκόσμιο επιστηστικό πρόγραμμα. Και αν μπορούμε να βρούμε ένα ή δύο εκατομμύρια για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τουλάχιστον την υποστήριξη που οι πληθυσμοί αυτοί θα μπορούσαν να λάβουν σε αυτό το επίπεδο. Επίσης ήθελα να σχολιάσω την ε, στάση που υπόθηκε και σήμερα ότι δεν υπάρχει καμία συμβολή στην δυνητική ανοικοδόμηση αν δεν υπάρχει ε, η προοπτική να μην καταστραφεί μέσα σε λίγες μέρες αυτό που έχουμε χρηματοδοτήσει όπως είδαμε στη Γάζα και ήταν πολύ λυπηρό. Τώρα για το κέρας της Αφρικής και τη Μιανμάρ. Οι αρχές μας φυσικά μας αναγκάζουν να δρούμε υπέρ των πληθυσμών ανεξάρτητα από την κατάσταση. Όμως υπάρχουν και οι ανθρωπιστικές κρίσεις που είναι ανθρωπογενείς και το Νότιο Σουδάν αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν σε αυτή την κατάσταση αν οι μανιακοί που το κυβερνούν αυτή τη στιγμή είχαν τα μυαλά στο κεφάλι τους. Ξέρω ότι δεν μπορούμε ως εκθαύματος να τα αλλάξουμε όλα αυτά, ούτε να πείσουμε την κυρία Σανσουκή την οποία σέβομαι. Δεν ήταν ποτέ στο Ολυμπιακό βάθρο που την είχαν άλλοι για μένα. Τώρα έχει την ε, ευκαιρία να φέρει ειρήνευση στη χώρα της και δεν το κάνει. Με όλη την πολιτική ισχύ που έχουμε, θα πρέπει να βοηθήσουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε, όμως ε, δεν πρέπει να βοηθάμε προσθέτοντας προβλήματα γιατί δεν χρησιμοποιούμε πολιτικές που θα έπρεπε. Τώρα, για τις μη αναγνωρισμένες χώρες. Είναι απλώς αόρατες, γιατί δεν μας επιτρέπεται να μπούμε. Θυμάμαι για τον Κάφκασο και για το Καραμπάχ, ε, όπου 100.000 άνθρωποι είχαν ε, αφανιστεί, βγήκαν στο δρόμο ε, λόγω των δεκαετιών πολέμου. το να μπούμε σε εταιρική σχέση με αυτή τη χώρα μας εμποδίζει από το να μπούμε εκεί σε αυτή την περιοχή. Δεν μπορούμε να μπούμε. Αν μας ενδιαφέρει η Ανατολική Ουκρανία και λογικό είναι αυτό, ίσως θα πρέπει να μοιαζόμαστε και για τους ανθρώπους ε, των οποίων τα χωριά δεν καταστρέφονται από τους ίδιους αλλά από άλλους ε, ανθρώπους πιο μοχτηρούς. Και για το Σομάλιλαντ ε, να πω ότι υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες ε, λόγω των αρχών της Σομαλιλάνδης, όμως τουλάχιστον υπάρχει μια αντιπροσωπεία που θα ανοίξει εκεί σύντομα και θα μπορούμε να έχουμε μια παρουσία για τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Ευχαριστώ. Μαρία Χόιμπουρκ, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ γιατί γρήγορα και αποτελεσματικά αντέδρασε στην ανθρωπιστική κρίση στην Αφρική. Είναι πολύ καλό να βλέπουμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια από την Ευρώπη είναι αξιόπιστη. Η Ευρώπη βέβαια μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερα εάν αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια ε, συμβάλλει περαιτέρω και στην ε, ανάπτυξη έχουμε εργαστεί σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε τη νέα ανακοίνωση για την δυνατότητα αντίστασης ως ε, μία από τις πρώτες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από, τις, από τα αποτελέσματα της αξιαλόγησης για την ανακοίνωση σχετικά με την επισητιστική ασφάλεια στην Αφρική βλέπουμε επίσης ότι αυτό όντως συμβαίνει. Στη συζήτηση με τους εργαζομένους στη δική σας γενική διεύθυνση φαίνεται ότι ε, υπάρχουν διάφορες ε, πτυχές ε, της δυνατότητας αντίστασης που δεν είναι πάντοτε αυτονόητες. Ας πούμε έχουμε οικογένειες, νοικοκυριά, το περιβάλλον. Είναι θέματα που δεν τα που τα παραγνωρίζουμε. Η ανθρωπιστική ε, κρίση στην Αφρική στην ουσία δείχνει πόσο σημαντική είναι η δυνατότητα αντίστασης ε, ως προς το περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ε, να έχουμε μία ε, γεωργική οικολογία η οποία θα προστεθεί στις δράσεις μας για να υποστηρίξουμε αυτή την δράση. Γιατί η γεωργική ε, οικολογία δεν είναι το ίδιο με την οικολογική γεωργία. Ε, η γεωργική οικολογία υποστηρίζει την έννοια ε, ε, ζώνες ε, που έχουν τη δυνατότητα μελλοντικά να φιλοξενήσουν μεθόδους καλλιέργειας που δεν θα συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος στην ουσία αυξάνουν την αντίσταση της περιοχής. Στη Γενική Διευθυνσιακό έχετε ασχοληθεί καθόλου με αυτή την γεωργική οικολογία ή με το ΦΑΟ, γιατί ο ΦΑΟ είναι σε αυτό το πρόγραμμα. Και το επιστηστικό πρόγραμμα στην ουσία σε αυτό επικεντρώνεται. Και άλλη μια μικρή ερώτηση για τη Συρία. Είπατε ότι θα υπάρξει ε, πρώτα μια πολιτική λύση και μετά θα μπούμε για να βοηθήσουμε. Όμως υπάρχει δυνατότητα ή ένας ε, μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει να εργαστούμε συστηματικά με τον πληθυσμό έτσι ώστε να έχουμε τα ντοκουμέντα που θα μας βοηθήσουν μετά να παρέμβουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μαρία, ο κύριος Βέντερ. Ε, ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περιγράψατε την κατάσταση με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, ιδιαίτερα στα της Αφρικής. Όταν μιλήσουμε για το κέρας της Αφρικής, μιλάμε και για την Ιεμένη και ίσως και για τον Νότιο Σουδάν. Θα πρέπει όμως να δούμε τι γίνεται και στην Ουγκάντα, γιατί πάνω από ένα εκατομμύριο προσφύγων έχουν πάει στη χώρα αυτή και είναι ένα επιπλέον πρόβλημα Υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες επίσης. Ε, το ε, ένα από τα προβλήματα είναι η ανθεκτικότητα. Η ανθεκτικότητα είναι μία από τις πέντε δράσεις της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιμένουμε πάντα ένα έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντωμεταξύ έχουμε προετοιμάσει ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την ανθεκτικότητα. Υπογραμμίζουμε τη συμφωνία την σημασία συγγνώμη, του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και για τις φυσικές καταστροφές και για την αύξηση των δυνατοτήτων αντίδρασης. Μπορείτε να μας πείτε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το έγγραφο αυτό. Μπορείτε να μας πείτε πότε θα δημοσιευθεί. Και μια τελευταία ερώτηση. Ποια θα είναι τα κεντρικά σημεία του συγκεκριμένου εγγράφου. Ποια θα είναι λοιπόν τα βασικά σημεία του εγγράφου αυτού, γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας 1,6 δις πολίτες του κόσμου αυτού σε χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται σαν εύθραυστες. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω γιατί έσβησαν τα φώτα, δεν είναι η ερώτησή σας που το έκανε αυτό. Νόμπερτ. Πάει και αυτός. Αναφερθήκατε στην αηφόρο ενέργεια, ίσως γιατί δεν έχουμε ήλιο σήμερα. Ευχαριστώ Επίτροπε που είστε ανάμεσά μας σήμερα. Στην αρχή αναφερθήκατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό και στην εκλεκτή συνεργασία που έχει η Επιτροπή μας με τις υπηρεσίες σας. Είναι αλήθεια αυτό. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, εμείς πήραμε μέρος σε όλα τα βασικά θέματα που είχαν σχέση με την διάσκεψη για τη μείωση των φυσικών καταστροφών και θα συνεχίσουμε τον επόμενο μήνα. Λόγω της κατάστασης της τέσσερις αυτές χώρες, Σουδάν, Ιεμένη, Σομαλία και Νιγηρία, αυτό περιλαμβάνει την κατάσταση στο σύνολο επίσης της περιοχής της λίμνης Τσάντ και ειδικά για την Ιγυρία και για την περιοχή του Τσάντ έχει υπάρξει κάποια πρόοδος. Οι κοινές στρατιωτικές δυνάμεις είναι αρκετά επιτυχείς εκεί στη δράση τους και μπορεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου η επιρροή του Μπόκο Χαράμ να μειωθεί. Όταν είχαμε μία συνάντηση με τις κοινέ στρατιωτικέ δυνάμεις εκεί μας ρώτησαν αν στον τομέα των στρατιωτικών είμαστε επιτυχείς και αν ναι πρέπει η ανθρωπιστική βοήθεια και η ε, κατεπίγουσα βοήθεια φυσικά να δοθούν άμεσα γιατί αλλιώς χάνουμε το πλεονέκτημα που έχουμε. Πώς λοιπόν η αναπτυξιακή βοήθεια συγγνώμη και η ανθρωπιστική βοήθεια συνδυάζονται σε αυτές τις περιοχές και μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών, των τεσσάρων χωρών, ιδιαίτερα της Νιγηρίας, να γίνουν πιο υπεύθυνε και να εμπλακούν περισσότερο. Τελευταίο θέμα είναι η πολιτική των Ηνωμένων Εθνών με τον Τραμπ ή μετά τον Τραμπ, όπως θέλετε. Είπατε ότι πήρατε μέρος σε ε, διασκέψεις δωρητών ε, βλέπετε κάποιες αλλαγές στην πολιτική των ΗΠΑ στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ευχαριστώ, Νόρμπερτ. Η Τερέζα Χιμένεθ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λίντα. Και ευχαριστώ θερμά τον Επίτροπο που ήρθε για συζήτηση και μας έκανε μια τόσο εκτενή παρουσίαση. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την εμπλοκή του και τη δέσμευσή του υπέρ της βελτίωσης κατάστασης των παιδιών. Γιατί μας απασχολεί ιδιαίτερο στο θέμα αυτό και ήμουν πρόσφατα στο Λίβανο και θα πάω και στην κοιλάδα Μπεκά. Εκεί δεν είναι μεγάλη η καταβλισμή προσφύγων, αλλά είναι μικρή καταβλισμή, 2.000 ε, χωρητικότητες Εκεί όμως είναι πολλά προσφυγόπουλα και όταν ε, ρώτησα πάτε στο σχολείο, ναι, κάποια αντίσκηνα ε, λειτουργούν ως σχολεία. Τα περισσότερα όμως ε, μικρά παιδιά δεν πήγαιναν καν στο σχολείο γιατί έπρεπε να πουλάνε μπισκότα και μερικές φορές ακόμη και στην... Ε, και η παραμονή του στο αντίσκηνο του στοιχίζει. Πρέπει να, να πληρώνουν ακόμη και γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό όταν μιλούμε για την ανθρωπιστική βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και, όλη την, και την αναπτυξιακή βοήθεια και όταν συζητούμε με εκπροσώπους του Λιβάνου και είχαμε επαφέ ε, με πολλού πολιτικού ηθήνοντε, ε, με ξέρει τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν μιλούσαν για την Ευρώπη. Δεν ανέφεραν την Ευρώπη ω ε, παράγοντα για την επίλυση τη σύγκρουση. Μίλησαν για τη Ρωσία, για το Ιράν, για την Τουρκία, για την Σαουδική Αραβία, τι Ηνωμένε Πολιτείε εννοείται, για τη Συρία, αλλά παρέλειπαν τελείως στην Ευρώπη στις αναφορές. Και κρίμα, παρά τις τεράστιες προσπάθειες που κάνουμε, δεν μετράμε καθόλου στα μάτια τους ω σημαντικός παράγοντας στην περιοχή. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση και την εικόνα μας εκεί. Και μια σύντομη ερώτηση για τη Βενεζουέλα. Γίνεται κάτι και ανέ ναι, τι για τη Βενεζουέλα. Γιατί στη Βενεζουέλα ε, λαμβάνει η χώρα μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και βρίσκεται στο σε ενός εμφυλίου πολέμου η χώρα. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε για τον πληθυσμό της Βενεζουέλας. Να προστατεύσουμε τον άμαχο πληθυσμό σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση που διανύει η χώρα. Επίσης, εκπονώ μια έκθεση για το χώρο της κοινωνίας των πολιτών και τη συρρήκνωση της κοινωνίας των πολιτών σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Θα ήθελα λοιπόν, όταν εσείς επισκέφτεστε αυτές τις χώρες, έχετε την εντύπωση ότι έχει υποχωρήσει η δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, συρρυκνώνεται ο χώρος κοινωνίας των πολιτών ή εμποδίζεται στο έργο τους από τους κρατικούς φορείς. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, πώ μπορούμε εμεί να συμβάλλουμε για να διευρυνθεί ο χώρο τη κοινωνία των πολιτών και η δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Γιατί όντω οι ακτιβιστέ ε, των ε, πολιτικών δικαιωμάτων υφίστανται πολλέ φορέ επιθέσει. Πώ μπορούμε να του βοηθήσουμε, λοιπόν. Ευχαριστώ και τελευταία, αλλά εκλεκτή επίση η Σεσίλια Κέγκε. Ευχαριστώ Λίντα και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο που μας παρουσίασε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει και την οποία συνεχίζει και μάλιστα σε μια τόσο μεγάλη κλίμακα την ανθρωπιστική βοήθεια. Ξεκινώντας λοιπόν από την ανθρωπιστική βοήθεια για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα, να μειώσουμε τους κινδύνους που έχουν τα εύθραυστα τμήματα του πληθυσμού και από την άλλη να δημιουργήσουμε ένα δεσμό ανάμεσα στο ανθρωπιστικό κομμάτι και την ανάπτυξη. Πρώτον, για την ανθεκτικότητα. Μα είπατε τι εννοείται, αλλά εννοείται και την ενίσχυση των τοπικών θεσμών. Το είπα αυτό γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να το συνδέσουμε με την ανθρωπιστική πλευρά και την ανάπτυξη και να δούμε ακριβώς τι γίνεται με την κοινωνία των πολιτών έτσι ώστε να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στους εμπλεκομένους και να μπορέσουμε σε ένα έδαφος να διασφαλίσουμε την παρουσία των, της ε, βοήθειας. Αναφερθήκατε σε χώρες, 14 χώρες, υπάρχουν και άλλες χώρες που δεν είναι ορατές. Εγώ επιστρέφω στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, την Κεντρική Αφρική, όπου πολλές περιοχές βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Θα ήθελα να μάθω ποιες είναι οι χώρες της περιοχής των λιμνών, της κεντρικής Αφρικής, όπου εσείς θα κατευθύνετε τις παρεμβάσεις σας. Και στο ίδιο κεφάλαιο ένα αίτημα προς εσάς και όλους τους συναδέλφους τις τελευταίες ημέρες ήρθε ένα αίτημα από την περιοχή του Κασάη, στην Δημοκρατία του Κόγκο. Όπως σας έχω πει, εκεί έχουν γίνει πολλές σφαγές και οι πολίτες ζουν στο εσωτερικό των δασών, είναι εκτοπισμένοι, ε, δεν βρίσκουν τροφή και το αίτημα το οποίο έχει πέρα από την έρευνα της υπόθεσης είναι να υπάρξει βοήθεια κατεπίγουσα. Ε, τι σκοπεύετε να κάνετε για το Κασάι. Το αίτημα είναι ισχυρό γιατί ο πληθυσμός της περιοχής αυτής δεν ε, βγαίνει από φόβο από τις δασικές περιοχές. Τελευταία παρατήρηση που αφορά τις ΜΚΟ και την Ιταλία για την έρευνα και διάσωση. Πολλές γίνονται έρευνες και διασώσεις από τις ΜΚΟ και αυτό γίνεται χάρη στις διάφορες δωρεές τις οποίες λαμβάνουν. Δεν έχουν άλλες μορφές ε, ε, χρηματοδότησης και κατηγορούνται για έλλειψη διαφάνειας. Τι θα κάνετε λοιπόν για τις ΜΚΟ αυτές που ασχολούνται με την έρευνα και διάσωση, τα νότια σύνορα. Εσείς μιλήσατε για το ανατολικό κομμάτι της Μεσογείου, εγώ μιλάω για το νότιο. Ευχαριστώ. Είναι πολλές οι ερωτήσεις, Επίτροπε. Πολλά τα θέματα. Έχετε το λόγο. Θα περάσω στα ελληνικά για να γίνω πιο συγκεκριμένος και ακριβής. Να ξεκινήσω από τον αγαπητό μου φίλο Ενρίγκε και θέλω να σχολιάσω τρία πράγματα από αυτά που ανέφερε ο, ο Το πρώτο θέλω να σχολιάσω αυτό τα φύγας από, τις, από τα πίνεμα από τις δημοσκοπήσεις. Ε, μέσα σε αυτό το κλίμα που αφισβητείται το European Project πιστεύω ακράδαντα ότι τα ποσοστά στήριξης του Humanitarian Aid και του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, του Civil Protection Mechanism, είναι πέραν από τα αναμενόμενα, διότι ε, φαίνεται ότι στις δημοσκοπήσεις θέλουν οι πολίτες να στείλουν μήνυμα στην πολιτική ελίτ πολλές φορές και για, την, για τις αδυναμίες μας και τις ελλείψεις μας σε ό,τι αφορά το γενικό ευρωπαϊκό project. Και γι' αυτό, εάν τα συγκρίνουμε με άλλα ποσοστά στο ίδιο ευρωμαρόμετρο, θα δούμε ότι τα ποσοστά της ανθρωπιστικής βοήθειας και του Civil Protection Mechanism είναι πάρα πολύ ψηλά. Που σημαίνει ότι ε, πρέπει να τα αξιολογήσουμε ως τέτοια. νέο σχέδιο δράσης. και η αξιολόγηση των δεσμεύσεων από το World Humanitarian Summit. Ε, είναι σε εξέλιξη το, το report. Σε λίγες μέρες θα μπορέσετε να το έχετε στη διάθεσή σας και νομίζω ότι θα ήταν ε, ευχάριστο ενδεχομένως να το συζητήσουμε κιόλα εάν θέλετε είτε σε συναντήσεις κατηδίαν είτε και εδώ ακόμη στην Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμφωνώ απολύτω με τον Ενρίκη ότι πρέπει να έχουμε αυτές τις αξιολογήσεις για να ξέρουμε με συγκεκριμένο τρόπο πού πάμε. Να έχουμε συγκεκριμένα φίκαρς και να εκτιμούμε, να αξιολογούμε τον εαυτό μας εάν πάμε σε σωστή κατεύθυνση ή πάμε σε λάθος κατεύθυνση. Για το, για το International Humanitarian Law δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ε, για μένα είναι από τις σημαντικότερες προτεραιότητες And τη ε, τελευταία δεκαετία το violation του humanitarian law αυξήθηκε οι επιθέσεις εναντίον civilians, εναντίον νοσοκομείων στη Συρία, στο Αφγανιστάν και η, λίστα είναι πολύ μεγάλη και νομίζω ότι η ανθρωπιστική κοινότητα πρέπει να βρει λύσεις. Ε, όπως ξέρετε Υπήρχε μια συνάντηση, η 32η International Conference of the Red Cross and the Red Crescents, στην προσπάθεια to strengthen the compliance with international humanitarian law. Εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε και να κάνουμε follow-up σε αυτό το process, αλλά βλέπω να υπάρχουν ακόμα δυσκολίες στο να δημιουργηθεί αυτό που εμείς οι, ως ανθρωπιστική κοινότητα θέλουμε. Να φτάσουμε στο σημείο να καταδικάζουμε αυτούς τους ανθρώπους με έναν τρόπο κατηγορηματικό. Ε, μαζί με τη Φεντερίκα Μολγερίνη as Vice President and ε, τα εξτέλαν το EAS ε, προσπαθούμε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δούμε πώς θα οθήσουμε τα πράγματα έτσι ώστε να γίνεται σεβαστό το international humanitarian law. Δεν έχω κάτι πιο συγκεκριμένο να σας πω τώρα. Δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να σας διαβεβαιώσω αλλά θέλω να διαβεβαιώσω ότι και εγώ προσωπικά και η Φεντερίκα αλλά και όλες οι σερβίσες και η ΕΚΟ προσπαθούμε έτσι ώστε να βρούμε εκείνους τους τρόπους για να αναβαθμίσουμε τη διεθνή προσπάθεια για, την, το σεβασμό του International Humanitarian Law. Δεν είναι εύκολη υπόθεση μέσα σε νομικά πλαίσια αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ήδη και αυτή η προσπάθεια που έγινε από το Red Cross και Red Crescent δεν είχε την επιτυχεί την τελική κατάληξη που θα θέλαμε κι εμείς. Δείχνει τη δυσκολία του εγχειρήματο. Ενδίκη ανέφερε κάτι συγκεκριμένα για το Ιράν. Ξέρεις ότι έχω επισκεφθεί δύο φορές την, τη χώρα αυτή. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου ότι ε, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία γιατί η χώρα αυτή για πάρα πολλά χρόνια φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων από το Αφγανιστάν ε, και θα συμβάλλει και στην πολιτική σταθερότητα της χώρας αλλά την ίδια στιγμή και στην θέση της στη διεθνή κοινότητα. Ε, από πλευράς των Ιρανικών αρχών έχω ένα θετικό μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι θετική απέναντί μας γιατί σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας προσφέρουμε και έχουμε αυξήσει τη βοήθεια ξέρουν πολύ καλά όμως ότι ήδη έχει περάσει η ανάγκη σε development aid, σε αναπτυξιακή βοήθεια. Συζητάμε με τον Νέβεν Μίμιτσα το όλο πακέτο Ιράν-Αφγανιστάν και αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε μέσω του development aid να βοηθηθεί και το Αφγανιστάν και το Ιράν. Δεν είναι πλέον θέματα emergency δεν είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά και μόνο την ανθρωπιστική βοήθεια. Σε ό,τι αφορά το education, in emergencies, θα ευχαριστήσω πάλι για τη βοήθειά σας. Είναι γεγονός ότι έχουμε αύξηση έξι φορές, six times, από την αρχή του, του mandate μου. Θα συνεχίσουμε και σίγουρα θέλουμε και εδώ να κάνουμε μια αξιολόγηση on the ground, να ξέρουμε ακριβώς που πάει, αλλά η αξιολόγηση που μπορεί να γίνει εμπειρικά, σας λέω ότι μέχρι τώρα ε, από τις δικές μου επισκέψεις αλλά και από την εμπειρία της DG ECHO είναι ότι όντως η επίδραση αυτών των λεφτών μέσω του Education Emergency έχει περισσότερο impact από ό,τι αναμέναμε. Και για να συνδέσω αυτή την απάντηση με την ερώτηση της αγαπητής συναδέλφου ε, σε ό,τι αφορά την κοιλάδα Μπεκά η κοιλάδα Μπεκά ήταν από τις περιοχές που επισκέφθηκα ε, στην αρχή και με όθησαν για να αυξήσω τη βοήθεια για το Education Emergencies και θα πω ότι όταν επισκέφθηκα πρώτη φορά την κοιλάδα Μπεκά αρχές του 2015 τα παιδιά που ήταν out of school ήταν περίπου 80% και τώρα έχουν μειωθεί στο 50%. Και αυτό εξαιτίας κυρίως της νέας ιδέας, της νέας προσέγγισης για το non-formal education, για το informal education. Και ήταν μεγάλη ε, επιτυχία αυτό το πράγμα. Βέβαια, πολλά απαιτούνται να γίνουν, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που είναι εκτός του σχολείου. Είμαστε σε συνεργασία με την, με, το, με την Λιβανέζικη κυβέρνηση, με την κυβέρνηση του Λιβάνου και μάλιστα είχαμε ένα ε, working dinner με την Μογκερίνη και τον Πρωθυπουργό και τέσσερις πέντε υπουργού που εστιάσαμε τη συζήτηση πάνω στο education Emergency. Στον αγαπητό συνάδελφο Έγκερ, που μπορεί και παρακολουθεί τη συζήτηση και στα ελληνικά. Ε, Συμφωνώ απολύτω με την διαπίστωση ότι εκεί που μπορούμε και προσφέρουμε 3 μπίλιον στην Τουρκία για να έχουμε ένα αποτέλεσμα πολύ ικανοποιητικό κατά την άποψή μου και θα πρέπει να το πούμε θα πρέπει να βρούμε και αυτό το ποσό που έχεις αναφέρει έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές στην περιοχή του Καζιάντεπ έτσι ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες. Θα το δούμε με τα services και στη νέα μου επίσκεψη θα είμαι στην Τουρκία πάλι τον Ιούνιο και θα προσπαθήσω να δω πώς θα βελτιώσω την κατάσταση. Σε ευχαριστώ για την επισήμανση. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι οι, οι συγκρούσεις που, που είναι man-made είναι ντροπιαστικές. It's a shame και ειδικά η περίπτωση του Σάου Σουδάν έχει απόλυτο δίκιο και θυμάμαι την επίσκεψή μου όταν είχα πολύ έντονη συζήτηση και σύγκρουση και με τους δύο αυτούς ηγέτες οι οποίοι δυστυχώ έχουν φέρει την καταστροφή σε αυτή τη χώρα το, νέο, το νεότερο κράτος στον κόσμο. Θεωρώ ότι η ανθρωπιστική κοινότητα και η διεθνής κοινότητα πρέπει να βρει τρόπους για να αντιμετωπίσει την περίπτωση του Σάου Σουδάν. Είναι μια περίπτωση που είναι ντροπιαστική για όλους μας. Ε, εγώ θα επισκεφθώ την Ουκάντα για ένα συνέδριο που θα γίνει με τον Γενικό Γραμματέα, τον Αντώνιο Κουτέρες, και υπάρχει περίπτωση να κάνουμε μια επίσκεψη και με τον Φιλίππο Κράντι του UNHCR μαζί στην, στο Σάου Σουδάν. Περιμένουμε όμως να δούμε. Γιατί καμιά φορά οι επισκέψεις μας στους South Σουδάνα, από αυτούς εκλαμβάνονται ως στήριξη και στις δικές τους προσπάθειες για ειρήνη η οποία δεν υπάρχει. Νομίζω ότι πρέπει να αυξήσουμε την ένταση της φωνής για να του σταλεί συγκεκριμένο μήνυμα. Η δική μου θέση είναι ότι χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τους δύο ηγέτες. Και συμφωνώ απολύτως μαζί σου, γιατί το πρόβλημα επεκτείνεται σε όλη την περιοχή του, του χώρου Φάρφρικα. Και Γι' αυτό έχουμε αυξήσει και την ανθρωπιστική ε, βοήθεια στην περιοχή. Το θέμα του Ναγκόνο Καραμπάχ, your obsession. Ε, δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω καλά την περίπτωση. Ομολογώ ότι ε, είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζω. Μέχρι τώρα ως DG ECHO δεν, είχαμε, δεν έχουμε γραφείο εκεί. We don't have any representation there, I think. Εργαζόμαστε με βάση τις αρχές, μπορούμε να παρέμβουμε, αλλά θα το δούμε μαζί. Θα σας δώσουμε πληροφορίες για να μπορέσουμε να ε, βελτιώσουμε αυτό που κάνουμε επί τόπου. Συμφωνώ απολύτως με τη συνάδελφο για την ανάλυση που έγινε σε ό,τι αφορά την γεωργική οικολογία και την γεωργική οικονομία. Και πρέπει με την συνεργασία του ΦΑΟ και έχετε απόλυτο δίκαιο να βρούμε τρόπους για να αυξήσουμε τη βοήθεια έτσι ώστε να χτίσουμε resilience ειδικά στις περιοχές της Αφρικής. Ε, είναι ένα, μια μεγάλη πρόκληση ακριβώς και για τους development αλλά και για τους humanitarian actors. Και όπως το έχετε θέσει ενδεχομένως να είναι το πιο σημαντικό challenge για τον έξους μεταξύ development και ε, humanitarian. Ε, είναι καλά να το συζητήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια. Αντιλαμβάνομαι ότι έχεις πολλές γνώσεις σε αυτό το θέμα και για μια συνάντηση είτε στο Στρασβούργο είτε μαζί με τα σέρβισέ μου για να δούμε πιο πρακτικά αυτόν τον τρόπο αντίδρασής μας. Διότι ξέρεις καλύτερα το θέμα και το έχεις δει και στην Αφρική όπω είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη μα συνάντηση. Αλλά έχεις δίκιο ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο σημασία γιατί είναι part of our resilient approach. Τι θα κάνουμε στη Συρία μέχρι να φτάσει η ειρήνη. Θα πούμε απλώς ότι περιμένουμε την ειρήνη για να επενδύσουμε έτσι ώστε να κάνουμε το rebuilding της χώρας. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ με... και θα θυμίσω την προσπάθεια που κάναμε με την Φετερίκα Μοκερίνη για το Αλέπο. Ε, τα πράγματα inside Syria είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολλές φορές δύσκολα to reach besieged areas. And, ε, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υποσχεθώ κάτι που δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουν. Όμως, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, είτε μέσω του Education Emergencies, είτε μέσω των ανθρωπιστικών οργανώσεων, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βρούμε λύση για να φέρουμε βοήθεια σε όλες τις περιοχές εντός Συρίας. Τώρα, η επανοικοδόμηση της χώρας δεν είναι εύκολο project, σίγουρα. Νομίζω ότι χρειάζεται μια μεγάλη διεθνής προσπάθεια ε, και ειλικρινά πιστεύω ότι δεν μπορεί να αρχίσει τώρα σε αυτές τις συνθήκες. Αυτό που μπορεί να γίνει τώρα είναι να απαντούμε στις άμεσες ανθρωπιστικές ανάγκες. Και αυτό είναι και ο ρόλος μας ως ε, Όσο μπορούμε τα καταφέρνουμε με μεγάλες δυσκολίες αλλά έχουμε πετύχει ακόμα και με πολιτικό τρόπο behind the scene να βρούμε ανθρώπους να τους βοηθήσουμε οι οποίοι, οι οποίοι ήταν ε, under starvation ε, κάτω από πολύ μεγάλες δυσκολίες να βρουν απλό φαγητό για να επιβιώσουν. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, σας διακόπτω, γιατί εγώ πρέπει να φύγω, να προλάβω το τρένο μου. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πόγκα, τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος ε, αυτός θα ολοκληρώσει τη συνάντηση. Κύριε Πόγκα, παρακαλώ, ελάτε εδώ. Mm. Για τις ερωτήσεις του αγαπητού φίλου Βέντα, ε, την Ουκάντα την έχω ήδη επισκεφθεί. Έχω δει από πρώτο χέρι τα προβλήματα και σε ένα από τους μεγαλύτερους καταβλισμούς που δυστυχώς σε έξι μήνες ο προσφυγικός πληθυσμός έφτασε να είναι 200.000 άνθρωποι από το Σάουστοδα. Και ήταν απίστευτη εμπειρία το πόσο δραματική ήταν η αύξηση αυτού του πληθυσμού. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ειδική μνήα για την Ουκάντα και έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία και έχουμε ήδη ε, διανύμει ένα μεγάλο ποσό ακριβώς για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των προσφύγων μέσα στην Ουκάντα. Σε ό,τι αφορά το έγγραφο για το resilience, ε, ο δικός μας σκοπός και η δική μας φιλοδοξία για αυτό το communication on resilience ε, είναι πρώτα να να παράσχουμε μια ευρύτερη κατανόηση της έννοιας ε, της ε, ανθεκτικότητας, να ξανασκεφτούμε ικανοποιητικά σε μια ολιστική προσέγγιση ε, και εάν χρειάζονται νέα εργαλεία στο resilience approach. Ε, νομίζω ότι μέχρι τον Ιούνιο, until June, we will see this. Θα δούμε αυτή την ανακοίνωση για την ανθεκτικότητα. Θα ήταν καλό να το συζητήσουμε ακόμη γιατί θα είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο πάνω στο οποίο θα αξιολογήσουμε τις μέχρι τώρα προσπάθειές μας στο Resilience που ήταν πάρα πολύ σημαντικέ, αλλά οπωσδήποτε πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε και συμφωνώ απολύτως ότι η συνεργασία μας είναι άριστη και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ε, επιμένουμε στις τέσσερις περιοχές που έχουμε το Looming Family. Ε, σε ό,τι αφορά ειδικότερα και τις επισημάνσεις σου για το Lane και την Νιγηρία ε, είχα μια ιδιαίτερη συνεργασία με τον Υπουργό Εξωτερικών στο Oslo Conference ε, μάλιστα τις τελευταίες μέρες Είχαμε επίσκεψη και από την καινούργια Humanitarian Coordinator για να, ακριβώς, για να δούμε πώς συντονίζουμε τις προσπάθειές μας. Ε, έχω αποφασίσει να επισκεφθώ την Ιγυρία μάλλον τον Ιούλιο ακριβώς για να κοιτάξουμε on the ground την κατάσταση. Ε, συμφωνώ ότι χρειάζεται μια συνεργασία ιδιαίτερη ε, Humanitarian Development και των στρατιωτικών οι οποίοι ξέρουν την περιοχή καλύτερα από όλους. Ε, όταν είχα επισκεφθεί Τσάντ και Νίγηρα ε, είχα επαφές με ε, ηγεσία των στρατιωτευμάτων της περιοχής και είδα και εγώ μια βελτίωση σε ό,τι αφορά την Πόκο Χαράμ αλλά μετά από τις συναντήσεις και με την Humanitarian Coordinator από την Νιγηρία πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι η συνεργασία των Humanitarian με τον Development Actors. Αυτή θα είναι η βάση για να αντιμετωπιστεί in medium and long term the Boko Haram influence in the society there. Βάλετε μια εξαιρετική ερώτηση που αφορά το το τι περιμένουμε από το New Trump Administration. Τον τελευταίο τρίμηνο συμμετείχα σε πάρα πολλά συνέδρια διεθνή και συνάντησα συναδέλφους Αμερικανούς από το administration μέχρι τώρα δυστυχώς υπάρχει μια σάφια τι θα γίνει με τη συνέχιση της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας από πλευράς Αμερικανών. Κανείς μέχρι τώρα δεν μας έχει διαβεβαιώσει για το αν θα συνεχιστεί και πώς θα συνεχιστεί. Ε, προτίθεμαι να κάνω το συντομότερο μια επίσκεψη στην Ουάσιγκτον για να διευκρινίσω τα πράγματα διότι αντιλαμβάνεστε ότι εάν έχουμε μία σαφή μείωση της βοήθειας από πλευράς Αμερικανών αυτό θα επηρεάσει γενικότερα το όλο σύστημα ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό για όλο τον κόσμο. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι εάν θα γίνει αυτή η μείωση θα επηρεαστεί περισσότερο το development aid παρά το humanitarian aid. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Όμως δεν μπορεί να υποθεί τίποτα με ασφάλεια και ακρίβεια. Πάντως θεωρώ τον εαυτό μου ως υπεύθυνο να ασκήσει την πολιτική πίεση που χρειάζεται για να συνεχιστεί η μέχρι σήμερα βοήθεια των Αμερικανών σε, αυτό, σε αυτά τα δύο τόσο ευαίσθητα φίλτς παγκοσμίω. Και τον θεωρώ ως προσωπικό μου στίχημα να είμαι advocate σε αυτή την προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα, είναι όντως ένα θέμα που το παρακολουθούμε. Δύσκολο θέμα, γιατί άπτεται της κυριαρχίας ενός κράτους και είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρέμβουμε ως DG ECHO ε, δίχως να υπάρχει η έγκριση από πλευρά κυβέρνηση. Ε, από το Σεπτέμβριο έχουμε χορηγήσει στους Κάριτας ένα project ε, στο health και στο nutrition σε τέσσερες διαφορετικές περιοχές. Ε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι το access είναι πρόβλημα εξαιτία του ότι χρειάζεται η συνεργασία της κυβέρνησης. Είναι δύσκολο and very sensitive issue, ε, but... Είναι ευαίσθητο θέμα, αλλά... Χρειάζεται να γίνει απέτηση από πλευράς κυβέρνησης μέσω του UN System. Ε, διαφορετικά ε, είναι δύσκολο να γίνει άμεση άμεσο intervention από πλευράς ε, Είμαστε σε συνεργασία και βλέπουμε μαζί με την Φεντερίκα και τον ε, Νέβεν Μίμητσα το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Είναι στα υπόψη με όλες αυτές τις δυσκολίες που ήδη έχω προαναφέρει. Τι αφήσαμε στην ερώτηση της συναδέλφου για το resilience νομίζω έχω καλύψει το θέμα. Στο αίτημα για, το, για την περιοχή του Κόγκο Καζάι δεν υπάρχει αφιβολία ότι θα πρέπει να το δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Είναι μέρος ε, της ε, ε, ανθρωπιστικής μας ε, ε, υπευθυνότητας, είναι μέρος είναι καθήκον μας να δούμε και όπως έχετε περιγράψει την κατάσταση. Τώρα είναι εδώ και η, η director του και θα το δούμε ακριβώς όπως το έχετε περιγράψει. Έχετε θέσει ένα θέμα για τις ε, NGOs στην Ιταλία έρευνας και διάσωσης. Γνωρίζω κάποιους ισχυρισμούς από κάποιον εισαγγελέα σε ό,τι αφορά παράξενες διασυνδέσεις. Ε, όντως ε, είναι για μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά funds να πηγαίνει με ένα τρόπο transparent και accountable διότι διαχειριζόμαστε λεφτά των Ευρωπαίων πολιτών διαχειριζόμαστε λεφτά των European taxpayers γι' αυτό είμαστε πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα την ίδια στιγμή όμως έχουμε σοβαρά requirements για το ποιοι NGOs συμμετέχουν στο European Funding και θέλω να το τονίσω γι' αυτό ε, αλλά από την άλλη και αναφέρομαι και στην ερώτηση της συναδέλφου Χιμένες ε, θεωρούμε ότι το Civil Society και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο σε όλες μας τις προσπάθειες στο humanitarian field. Γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και από εσά οποιασδήποτε πληροφορίε ναι, για να προστατεύσουμε την προσπάθεια των μη κυβερνητικών οργανώσεων που βοηθούν τόσο πολύ on the ground. Σε ό,τι αφορά την, το Central African Republic, και τις μεγάλες λίμνες για φέτος η βοήθειά μας είναι περίπου 45 εκατομμύρια και έχετε απόλυτο δίκιο οι ανάγκες είναι τεράστιες. Αλλά με φέρνει και στην τελική μου κατάληξη για να ενισχύσω αυτό που είπα πριν για το Trump Administration εάν δυστυχώς έχουμε μια μείωση της βοήθειας που προσφέρεται από αμερικάνικης πλευράς είτε στο humanitarian aid είτε στο development aid αντιλαμβάνεστε ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι από μόνοι μας δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις μεγάλες απαιτήσει που η ίδια η ζωή και οι ίδιες οι κρίσεις ήδη αναδεικνύουν καθημερινά. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει ναι και είπα και πριν ότι θεωρώ ότι ένας από τους δικούς μου ρόλους προσωπικά ως Commissioner for Humanitarian Aid να ασκήσουμε πολιτική πίεση για να μην μειωθεί η βοήθεια που μέχρι τώρα ισορροπούσε τη συνολική βοήθεια από πλευράς Αμερικανών. Είναι μεγάλης σημασίας να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικανών σε ό,τι αφορά το development και το humanitarian aid. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για αυτή την τόσο γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση. Κάθε φορά που έρχομαι στην, στο DEVE Committee σας ομολογώ ότι και μαθαίνω και κερδίζω και από τις δικές σας ευαισθησίες και από τις δικές σας εισηγήσεις. Ευχαριστώ πολύ και το γραφείο μου είναι πάντα ανοιχτό για μια προσωπική συνάντηση και συζήτηση για όλα τα θέματα. Merci, Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Εκ μέρου τη Επιτροπή μα, τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά για τι απαντήσει που δώσατε στις ερωτήσεις ε, των συναδέλφων και σας ευχαριστούμε θερμά επίσης για την στενή μας συνεργασία και σας ευχόμαστε καλό κουράγιο για τη συνέχεια. Χαίρετε. Nous arrivons στο τέλος των εργασιών μας. Ε, το πρώτο τελευταίο σημείο, τα διάφορα. Υπάρχουν ε, θέματα για τα διάφορα. Όχι θαυμάσια. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα γίνει στις 29 Μαΐου 2017, 3 με 6.30 και 30 Μαΐου 9 με 10 και μισή. Ή 12 και μισή μάλλον. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς και να κηρύξω το πέρα στη συνεδρίαση. Merci beaucoup. Σα πω